Λοιπόν, τέταρτη ή πέμπτη δοκιμή τώρα. Η γνωμοδότηση την οποία πρόκειται να συζητήσουμε σήμερα, η γνωμοδότηση αυτή ε, θα υποβληθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία Επιτροπή Περιβάλλοντος θα τοποθετηθεί στην πρόταση που υπάρχει να αλλάξει η περιεκτικότητα θείου σε κάψιμα πλοίων. Οι αλλαγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγούν στο να συγχρονιστεί η οδηγία με τις ε, τροπολογίες και το παράρτημα το οποίο έχει εκδώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο IMO. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Παρότι οι έξι, τα έξι αυτά παραρτήματα εγκρίθηκαν ήδη το 2008, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της για αλλαγή της οδηγίας μόλις πριν από λίγους μήνες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ορισμένες από τις ε, πιο αυστηρές προϋποθέσεις, αυστηρούς όρους για τα καύσιμα των πλοίων ετέθησαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2010 ε, και όσα δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Ιούλιο του 10 ε, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Πρώτη του 12. Υποθέτω λοιπόν ότι είχαν ήδη προϋπάρξει κάποιες συζητήσεις μέχρι το 2008 και οι συζητήσεις αυτές αφορούσαν επίσης ε, τη γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων επιτροπών. Αυτά λοιπόν ε, έλαβαν τελική μορφή σε μια κοινή γνωμοδότηση όπου καθίσταται σαφές ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ε, καθαρότητα του αέρα και κατέστη επίσης σαφές ότι η ε, ρήπανση που προέρχεται από τα πλοία είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πηγή ρήπανσης. Υπάρχουν δύο χώρες οι οποίες ε, δεν έχουν επικυρώσει τους όρους, η Εστονία και η Λετωνία. Βέβαια δεν είμαι σίγουρη για το κατά πόσον ε, τα απορθμία μεταξύ Εστονίας και Φινλανδίας ε, πρέπει να καλύπτουν τους όρους ή όχι. Τώρα λοιπόν που τελειώνουν, εκπνέουν οι προθεσμίες. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε, ξέρετε, δυστυχώς εμείς δεν είχαμε καταλάβει ε, περί τίνος πρόκειται. Αν ήμασταν λαϊκιστές ε, θα λέγαμε, α, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, κρίμα και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει η συμπεριφορά μας ε, να προσαρμοστεί και να προχωρήσουμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε ψηφίσει. Γιατί σε τελική ανάλυση εμείς επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στους ε, διεθνείς ε, οργανισμούς. Οι κανονισμοί ε, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Έτσι και αλλιώ πρόκειται μέχρι το τέλος του έτους να τεθούν σε ισχύ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ε, προτείνω ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε την αναβολή των νέων αυτών κανονισμών. Όσον αφορά στο παράρτημα υπαριθμών 4. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη οφείλουν να μην πιέζουν τις εταιρείε εκείνες οι οποίε καταβάλουν πραγματικέ και σοβαρέ προσπάθειες για να προσαρμοστούν στου ε, κανονισμούς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξή. Η περιεκτικότητα σε θείο η μείωση τη περιεκτικότητα σε θείο έχει ω στόχο τη βελτίωση της ατμόσφαιρας. Ο κανόνας αυτός ε, πρέπει να ισχύει για όλες τις ε, θάλασσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πρωτοπόρα στην κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει άλλη λύση. Η τροπολογία μου υπαριθμών 2 ε, είναι συναφής με αυτά που σας είπα μόλις τώρα. Πάμε στο τρίτο οι αυξημένες τιμές των ε, καυσίμων πλοίων μπορούν να επηρεάσουν ε, τις ε, εμπορευματικές συνδυασμένες μεταφορές και γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα πρέπει εδώ να παίξουν ρόλο και οι θαλάσσιες μεταφορές. Η έρευνα που γίνεται είναι αμφιλεγόμενοι. Μερικοί λένε ότι πράγματι υπάρξει επιρροή των εμπορευματικών μεταφορών, άλλοι πάλι λένε όχι. Κατόπιν, εγώ δεν προτείνω την πρόταση, δεν στηρίζω την πρόταση Κομισιόν να απαγορευτούν, απαγορευτούν πλήρως καύσιμα με περιεκτικότητα θείου πάνω από 3,5%. Επίσης, προτείνω αυτό να ισχύει μόνο για καύσιμα που χρησιμοποιούν τα πλοία και όχι καύσιμα που μεταφέρουν τα πλοία. Επίσης, όσον αφορά το ε, υγροποιημένο αέριο, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, μετά από ε, κάποια χρόνια δεν θα πρέπει να έχουμε αγνοήσει την δημόσια υγεία και γι' αυτό εγώ ε, προτείνω αυστηρότερους ε, κανονισμούς και σε άλλες θάλασσες και για τα επιβατηγά πλοία. Όχι μόνο εκείνα τα οποία εκτελούν τακτικές ε, διαδρομές. Αναφέρομαι στις ανθρωπολογίες υπαριθμών 8 και 9. Και κατόπιν επιθυμούμε να έχουμε και μία έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς ακριβώς ε, συνεχίζεται η εφαρμογή των κανονισμών, αν έχει περιοριστεί η ρήπανση και να ενημερωθούμε και για το κατά πόσο χρειάζονται νέες νομοθετικές προτάσεις ε, κατά όσο το ζητάει αυτό η Επιτροπή. Αναφέρουμε στην τροπολογία ε, υπαρθμών 10. Εσείς υποβάλλετε 101 τροπολογίες και από κοινού με τον εισηγητή προσπάθησα να προτείνω συμβαστικές προτάσεις Όσον αφορά την πρόσβαση σε χρήση εναλλακτικών ε, καυσίμων, των πλυντρίδων και άλλα, ε, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε και ε, τον δρόμο της ε, κύρωσης. Τροπολογία υπαριθμών C. Βαστική γάμα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προτάσεις ε, για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ε, οικονομικές δυσκολίες. Πάμε στην συμβαστική πρόταση ΔΕΛΤΑ. Αυτή αφορά το υγροποιημένο αέριο και την ασφάλεια στη θάλασσα, τη σχετική σύμβαση. Επίσης, υπέβαλα και την συμβαστική πρόταση Ι, e, η οποία αναφέρεται σε άλλα καύσιμα ε, και σε άλλες χημικές ουσίες όπως είναι ο άνθρακας. Εγώ δεν στηρίζω αυτή τη συμβαστική πρόταση, όμως κατά την άποψή μου τελικά αυτή η συμβαστική πρόταση ε, θα μπει στην αιτιολογική σκέψη και όχι στο κύριο σώμα της οδηγίας. Εγώ ως εισηγήτρια δεν στηρίζω αυτή τη συμβαστική πρόταση, αλλά βεβαίω ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τη στηρίξουν οι συνάδελφοι. Με βάση αυτά τα οποία είπα μέχρι τώρα και, τις, ε, και την αιτιολογική σκέψη, βλέπετε στον κατάλογο ε, ψήφου ποια ακριβώς είναι η θέση μου και η θέση δική μου απορρέει από την τελική σκέψη. Ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σας ε, για σχόλια. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Ήταλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια για την ε, τόσο πολλή δουλειά που έκανε. Η συνεργασία μας ήταν γενικά πολύ καλή. Θα μπορούσα να υποστηρίξω από την ομάδα μου πολλές από αυτές τις τροπολογίες και τις συμβαστικές. Για την πρώτη συμβιβαστική εμείς ε, αφήνουμε κατά συνείδηση ψήφο. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Εγώ εκπροσωπώ την Φιλανδία, οπότε από πλευράς της Φιλανδίας η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα ατυχής. Το 2008 ξεκίνησε η απόφαση αυτή. Είναι πάντως αλήθεια ότι το 2008 ο κόσμος ήταν εντελώ διαφορετικός από ό,τι σήμερα. Και οι αξιολογήσεις για το περιβάλλον που είχαν γίνει τότε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ήταν επίσης κάτι το εντελώ διαφορετικό. Βέβαια, στην πολιτική ξέρω ότι ποτέ δεν αναγνωρίζονται τα σφάλματα και αυτό είναι το πρόβλημα. Ήδη πριν από ένα χρόνο είχαμε πει ότι αν στις μεταφορές οι αποφάσεις για τις εκπομπές λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα τμήμα της μόνο. Καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως προχωράμε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο μας, μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Και για τη Φιλανδία όλος ιδιαίτερος. Σας δίνω το παράδειγμα της Φιλανδίας, αλλά Βλέπετε και η Ρωσία, παρόλο που έχει υπογράψει, δεν θα χρησιμοποιήσει την νέα συμφωνία. Θα σταθεί στις παλιές εκπομπές, στα παλιά όρια. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν είναι καλή ιδέα να αντιμετωπίζουμε μερικές μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν, πιστεύω, πιο λογικό να καθυστερήσουμε την απόφαση περισσότερο. Πάντως, για τις συμβαστικές τροπολογίες, νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Και ελπίζω, ελπίζω οι υπόλοιπε τροπολογίες πέρα από την τελευταία να περάσουν και να έχουμε μια αξιοπρεπή λύση. Ο κύριος Ζέμκε από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω εγώ ευχαριστώντας την εισηγήτριά μας για την δουλειά που έχει κάνει. Εκ μέρους της δικιάς μου πολιτικής ομάδας, εκ μέρους δηλαδή των σοσιαλιστών και δημοκρατών, θέλω να σας ε, μεταφέρω διάφορα σχόλια. Γνώμη μας είναι πως είναι αναγκαίο η οδηγία αυτή να εγκριθεί. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό ξανά και ξανά, γιατί εγώ έχω δουλέψει πάνω στην οδηγία αυτή και ξέρω ότι έχουν ακουστεί πολλές διαφορετικές φωνές και απόψεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα επιχειρήματα. Γιατί από τη μια μεριά έχουμε προφανή επιχειρήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος, τόσο της θάλασσας, των λιμανιών, σου και του αέρα. Από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά, ως Επιτροπή Μεταφορών, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και όσον αφορά τις εξελίξεις τις μεταφορές. Άρα και τις θαλάσσιες μεταφορές. Συνεπώς, πρέπει να καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες να είναι τέτοιες ώστε να υποφωλείται και το περιβάλλον, αλλά από την άλλη μεριά να μην οδηγούν και σε μια κατάσταση όπου καταστρέφονται μεταφορές σε ορισμένες χώρες μέλη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι η οδηγία αυτή είναι καλή. Την έχουμε δουλέψει σε βάθος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να σας μιλήσω τώρα για τις συμβαστικές τροπολογίες. Θέλουμε να στηρίξουμε και τις πέντε συμβαστικές τροπολογίες που προτείνονται. Η άποψή μας είναι πως είναι λογικές, καλές και επίσης πιστεύουμε ότι η οδηγία αυτή πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια, όλα δηλαδή τα ύδατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις συμβαστικές τροπολογίες θα έλεγα ότι πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω πάνω στην γάμα. Εκεί υπάρχει κάπως διαφορετική άποψη στην ομάδα μου σε σχέση με την εισηγήτρια όπως και με τη συμβαστική τροπολογία ε. Γιατί η ουσία της ε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει νέες προτάσεις για το θείο, χωρίς όμως να λέμε ποιο πρέπει να είναι το χρονοδιάγραμμα ή το χρονικό όριο και λέμε ότι δεν είναι πολύ σημαντικό όταν πρόκειται για την ποιότητα των καυσίμων ή του περιβάλλοντος όμως έτσι. Από τις 120 πάντως τροπολογίες και στην πολιτική μας ομάδα αλλά και με τις άλλες πολιτικές ομάδες έχουμε συζητήσει και συμφωνούμε λίγο πολύ. Το πρόβλημα είναι τροπολογία 65. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει μεταξύ μας ξανά και ξανά όπου ο κύριος Τσίλε προτείνει να εισαγάγει πολύ αυστηρές λύσεις. Αντί για το 3,5% δηλαδή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκείνος προτείνει 1,5%. Αυτό είναι κάτι επίμαχο, ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα και σίγουρα θα χρειαστεί να ζητήσουμε την άποψη ειδικών και αύριο το πρωί θα έχουμε καταλήξει πώς θα τοποθετηθούμε ως πολιτική ομάδα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και το, την εισηγήτρια. Υπάρχουν πολλές και διάφορες τροπολογίες που έχουμε υποβάλει και εμείς. Πιστεύουμε ότι η γραμμή που έχει επιλέξει η εισηγήτρια είναι σωστή γιατί όντω έχει μια σωστή οπτική γωνία. Φυσικά και υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι δυσαρεστημένες. Το καταλαβαίνουμε αυτό και καταλαβαίνουμε και την επιχειρηματολογία τους, αλλά από την άλλη μεριά όλες οι χώρες πλήττονται λίγο πολύ. Και όλες θα έχουν κάποιες αρνητικές συνέπειες από μια τέτοια ρύθμιση. Πάντως, Υπάρχουν χώρες που τώρα είναι έτοιμες και άλλες που δεν είναι έτοιμες. Αυτές που δεν είναι έτοιμες δεν μπορεί η κροκοδίλια δάκρυα τώρα να χύνουν και να λένε ότι α, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει επίσης να καλύπτει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε. Είχαμε μιλήσει για τρεις περιοχές, αλλά θα έπρεπε να καλύπτονται και άλλες. Ο ανταγωνισμός πρέπει να βάζει όλες τις περιοχές επί ίσης ώρες. Το ίδιο έχω να πω και για τις άλλες συμβαστικές τροπολογίες. Την α δεν θα τη στηρίξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι εκτός πεδίου συζήτησης. Κατά τα άλλα, θα ακολουθήσουμε τη γραμμή της εισηγήτριας. Η αγγλική αντιπροσωπεία πάντως από την ομάδα μας ε, έχει πει ότι θα ψηφίσει διαφορετικά. Κατά τα άλλα, σας είπα. Ευχαριστώ πολύ. δεν θα σχολιάσω, θα το αποφύγω. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να σας πω ε, ένα ευχαριστώ ε, στην εισηγήτρια εκ μέρους των ε, Πρασίνων και θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στην ίδια την έκθεση. Υπάρχει το εξής ερώτημα δεν θα έπρεπε να ενδιαφερόμεθα για το κατά πόσον θα περιορίσουμε την περιεκτικότητα σε θείο. Αυτό ήδη ορίζεται από το Μάρπλ, ε, το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ε, τηρούμε. Όσον αφορά τώρα την ομάδα των πρασίνων, εγώ έχω καταθέσει 20 περίπου τροπολογίες ε, αλλά θα ήθελα να μιλήσω πολύ σύντομα για τις ε, συμβαστικές. Συμφωνούμε απόλυτα με τη συμβαστική Α και εμείς ε, θεωρούμε, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να επεκταθούν οι ΠΕΘΑ. Όσον αφορά την συμβαστική Β, είχαμε μια μακρά συζήτηση στη συνεδρίαση των σκιωδών και ήλπιζα ότι αυτό θα καταλήξει σε επικοδομητικές παρατηρήσεις. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Κατόπιν τούτου δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη συμβαστική τροπολογία και γι' αυτό θα ήθελα το δικό μας το όνομα να αφαιρεθεί από αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Όσον αφορά ε, την τρία, ε, δεν πιστεύουμε ότι αυτό που αναφέρεται ως συνέπεια θα προκύψει απαραίτητα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η μείωση η, η ε, μεταφορά σε οδικές μεταφορές θα γίνει σε άλλα επίπεδα. Άρα δεν θα έχουμε εδώ σημαντικές επιπτώσεις. Ούτε συμφωνώ με αυτό που αναφέρεται ότι η κονδύλια από το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο ή το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτό το στόχο. Άρα δηλαδή ε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη συμβαστική σε ε, πράγματι όλοι οι τρόποι μεταφορών θα πρέπει να προσπαθήσουν να απορροφήσουν το εξωτερικό κόστος και αυτό ε, δεν μπορεί να είναι ε, η εξαίρεση για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Τώρα, πολύ καλά νέα όσον αφορά το υγροποιημένο αέριο. Αυτό, κατά την απόψή μας, πράγματι έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κλασικά παραδοσιακά καύσιμα και θέλουμε να ενθαρρύνουμε ε, την χρήση του υγροποιημένου αερίου. Εδώ θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια από το πρόγραμμα Μαρκο Πόλο. Αυτό δηλαδή που θα γίνει τελικά πρόεδρε είναι εμείς θα ζητήσουμε ψηφοφορία κατά τμήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη μετάβαση ε, προς το υγροποιημένο αέριο αλλά σας λέω όχι με τη χρήση των κονδυλίων από το πρόγραμμα Μαρκο Πόλο. Και τέλος, ως πράσινη να σας πούμε επίσης ότι με μεγάλη μας χαρά να στηρίξουμε τη σημαστική πρόταση Ι. E. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη συζήτηση που έχει προκύψει συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν βέβαια ε, διαφορετικές οριακές τιμές ε, του θείου στις ελεγχόμενες περιοχές, στις περίφημες πέθα, αλλά και μέσα στις δικές μας τις πολιτικές ομάδες. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Αυτά λοιπόν σίγουρα έχουν σχέση και με τα εκάστοτε εθνικά οικονομικά συμφέροντα. Αυτό δεν πρέπει να το απορρίπτουμε. Ρίχνοντα μια ματιά στη Φινλανδία, γνωρίζω ότι υπάρχουν στη χώρα αυτή πολύ μεγάλοι φόβοι για το πώ θα προστατεύσει τον τομέα τη ξυλία τη και την αυτιλία τη. Όσον αφορά τώρα ε, τις ε, θαλάσσιες μεταφορές μικράν, μικρών αποστάσεων υπάρχουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στο κόστος των καυσίμων. Αν λοιπόν κάνουμε την αξιολόγηση θα δούμε ότι 60% έχουν αυξηθεί τα κάψιμα σε αυτές τις ε, μικρές μεταφορές ή θα αυξηθούν εάν τελικά επιτρέπεται θείο στα πλοία, με, αν επιτρέπονται καύσιμα στα πλοία, με περιεκτικότητα μόνο 0,1% θείο. Άρα δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογηθεί η στρατηγική μας για το μέλλον, κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί η μετάβαση από ε, τις οδικές μεταφορές ε, στις θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει να δούμε μήπως ακολουθούμε λάθος κατεύθυνση. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας μόνο τρία χρόνια. Ε, είχαμε διάφορες ακροάσεις για το ποιες τεχνικές δυνατότητες υφίστανται για να μπορούμε να παρέμβουμε. Αναμφισβήτητα το υγροποιημένο αέριο είναι πρόσδεκτο, φιλικό προς το περιβάλλον, με χαμηλή περιεκτικότητα θείου. Ε, θα πρέπει όμως μέχρι τότε, μέχρι να χρησιμοποιείται βρέως, να έχουμε κατασκευάσει και τις μονάδες ανεφοδιασμού. Αυτό ε, δεν ισχύει. Ή οι πλυντρίδες ε, βρίσκονται εν τη γενέση τους. Επίσης ε, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξοπλίσουμε το στόλο. Γι' αυτό λοιπόν η τροπολογία μου, η Παρτμόν 16, ε, λέω εκεί οι ε, μεταφορές μικρών αποστάσεων να λάβουν μία μεταβατική περίοδο 5 ετών και στις, στα μεγάλα τα σκάφη ε, ανοιχτή θαλάσσης. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κόστος είναι κατά κανόνα γύρω στο 2% τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα κράτη αυτά είναι εκείνα που έχουν τις ε, διαπραγματεύσεις με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς απλά εφαρμόζουμε αυτά που αποφασίζονται. Γι' αυτό λοιπόν τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα πρέπει να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έτσι ώστε να βρούμε μια πρακτική και εφαρμόσιμη λύση και να μην αδειάσουμε το μωρό μαζί με τα απόνερα. Έχω άλλους πέντε ομιλητές, συν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Φλέκενστάιν έχει το λόγο. jetzt. Herr Vorsitzender, ich würde gerne der Berichterstatter... Κοιτάξτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πάρα πολύ καλή δουλειά της, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει φτάσει πια η στιγμή να κάνουμε κάτι που να αφορά τη θάλασσα. Δεύτερον, καθίσταται σαφές ότι αυτά πρέπει να λάβουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι σε μεμονωμένα τμήματα της Ευρώπης. Τρίτον, από ό,τι φαίνεται χρειαζόμαστε και μία φάση προσαρμογής. Ο κύριος Κούν επισήμανε ότι ε, χρειαζόμαστε και κονδύλια για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Τέταρτο, και προτελευταίο, δεν είμαι σίγουρος ε, για το κατά πόσον οι επενδύσεις ε, στο υγροποιημένο αέριο ε, θα μας βοηθήσουν. Πριν από 35 χρόνια, όταν άρχισα να εργάζομαι σε έναν όμιλο επιχειρήσεων που ασχολιόταν με το αέριο, μου είπαν τότε θα υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο, το υγροποιημένο αέριο. Μα έχουν περάσει 35 χρόνια και δεν έχουμε προχωρήσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το υγροποιημένο αέριο δεν είναι παλάτια στην άμμο, είναι κάτι συγκεκριμένο που να μπορεί κανεί να το προχωρήσει. Πάω στη δική μου την τροπολογία, την 53. Ε, Βεβαίω και με ενδιαφέρει να καταστήσουμε σαφέ ότι μα είναι παντελώ αδιάφορο ε, το πώ ε, κινούνται τα πλοία. Αν θέλετε, α βάζουν μόνο θείο. Εμά δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτό που μα νοιάζει είναι τι βγαίνει πάνω από την καμινάδα του. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με την κυρία Μάσινερ, όπου βέβαια στη δική μου την τροπολογία τη βρίσκω πολύ καλύτερη. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Θα ακούσουμε τώρα την άποψη της κυρίας Μάισνερ. Από ό,τι φαίνεται ο προλαλής και εγώ και οι δυο μας ασχολούμαστε με πολιτική που αφορά τη θάλασσα. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τώρα κράτη-μέλη, ήταν βέβαια γνωστό αυτό, ε, κράτη-μέλη ε, που έχουν υπογράψει αυτές τις συμβάσεις στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Πρέπει όμως να αλλάξει το πρότυπο. Να έχουμε τώρα μια συνδυασμένη λύση, ακριβώς αυτό που προτείνει η συγγήτριά μας. Δηλαδή, αφενός να στηρίξουμε να προχωρήσει το υγροποιημένο αέριο. Εγώ διαφωνώ με αυτά που λέξαμε μέχρι τώρα. Στο Ρότερνταμ, παρήματο χάρη, υπάρχουν πάρα πολλέ δυνατότητε ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο. Μέχρι το 2015 θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα μπορούμε να προσφέρουμε την υποδομή. Είναι η εναλλακτική λύση. Πλυντρίδε. Εδώ υπάρχουν πολλέ δυνατότητε. Η τεχνολογία δεν έχει εξαντληθεί και θα δούμε τι θα γίνει. Και κάτι καινούριο. Από του φιλελεύθερου ακούσαμε, είχαμε ένα ε, σεμινάριο ε, και την ίδια μέρα είχαμε και ένα άλλο σεμινάριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τις πλυντρίδες και αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν μια εισηγήτρια από τις ΗΠΑ που είπε ότι στις ΗΠΑ εν μέρη προαιρετικά έχουν εισάγει ε, αυστηρότερες οριακές τιμές και όπου υπήρξαν ουσιαστικές παραβάσεις εκεί επιβλήθησαν κυρώσεις. Και αυτό συνέβη μετά την κατάθεση των δικών μας των τροπολογιών. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που η συγγήτρια δίνει πιο αυστηρό ύφο σε αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Εγώ θεωρώ ότι αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγα σημεία. Ο κ. Βαντάλεν έτσι και αλλιώς κάλυψε διάφορες περιπτώσεις είναι σαφές ότι θα υπάρξει και εδώ μια συμφωνία. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε ότι κάθε μορφή μεταφοράς πρέπει να είναι το μέγιστον καθαρή. Και θα πρέπει να πάρουμε μέτρα γι' αυτό ακριβώς το στόχο. Από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Φοβάμαι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο μεταφοράς, είτε το θέλουμε είτε όχι αναγκαστικά θα δούμε μια μεγάλη αύξηση στο κόστος της ναυσιπλοείας όταν θελήσουμε να διευρύνουμε τα μέτρα αυτά νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν άκερο και σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα μπορούσαμε να το προτείνουμε και να το στηρίξουμε. Νομίζω ότι το όριο είναι αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και το IMO. Αν υπάρξει μια συμφωνία και στο IMO, οι χώρες δηλαδή που συμμετέχουν στον διεθνή αυτό οργανισμό, πέραν τούτου δεν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να συζητάμε κάποια θέματα, αλλά να μην αγνοούμε παρακαλώ τι θέλει η διεθνής κοινότης. σχετικά τώρα με τα πλοία τα οποία εκφεύγουν του Ίκας. Αυτό έτσι και αλλιώς θα συμβεί το 2020. Γιατί να προσπαθήσουμε αυτό να το κάνουμε πιο πρόωρα, Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο. Για τη διαθεσιμότητα του καυσίμου προφανώς θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα αυτή και γι' αυτό και υποστηρίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία Β αυτός είναι ο στόχος. Συμφωνούμε με την συμβιβαστική αυτή πρόταση. Και εφόσον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ρευστοποιημένο ή το υγροποιημένο φυσικό επίσης αέριο και αυτό εφόσον μπορεί να γίνει, γιατί όχι. Πέραν αυτού όμως τίποτα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει καταληκτικά θα έλεγα ότι η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να μην καταδικάσουμε σε πτώχευση τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γιατί αυτά τα οποία λέγουν ορισμένοι εκεί μας οδηγούν. Λοιπόν, ναι, πρέπει να είμαστε όσο πιο καθαροί γίνεται, αλλά παρόλα αυτά με ρεαλισμό πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Θέλουμε να μειώνουμε τις οδικές μεταφορές, ε, γιατί όχι φυσικά, αλλά ε, προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς ε, χρησιμοποιώντας καλύτερα τις θαλάσσιες μεταφορές και τις παραποτάμιες μεταφορές επίσης. Ας το κάνουμε αυτό σεβόμενοι τις διεθνείς συμφωνίες, την διεθνή κοινότητα. Αν το κάνουμε αυτό τότε θα πετύχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, αγαστή συνεργασία ε, κοιτάξτε, εγώ είμαι 7 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε μιλήσει πολύ συχνά για τις ε, εκπομπές ε, στη θάλασσα. Και λέμε, εμεί τα θέλαμε, αλλά δεν θέλει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Να τώρα που θέλει και τώρα τι λέμε εμείς. Α, ωραία, θέλετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν είναι σωστό αυτό. Αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την κατάσταση με τις εκπομπές, είτε από τα αεροπλάνα είτε από τα αυτοκίνητα είτε οπουδήποτε αλλού. Ε, θα πρέπει να είμαστε πιο συνετοί γιατί πολλοί λένε θα αυξηθεί το κόστος και τελικά όλα θα μεταφορθούν ε, στις αντικές μεταφορές. Μόνο που όταν μιλάμε για τους σιδηρόδρομους, ε, τελικά τι κάνουμε, ε, αυξάνουμε το κόστος, πάνε όλες οι οδικές μεταφορές και δεν κάνουμε τίποτα. Μιλάμε μόνο για εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστος και τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και στον κόσμο μεταφέρονται πάρα πολλές ανοησίες, ε, πράγματα που είναι πολύ φτηνά, που ε, ρηπαίνουν το ε, περιβάλλον γιατί όσον αφορά τη θάλασσα, εκεί υπάρχουν ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις και εφόσον υπάρχουν αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, θα πρέπει οι θαλάσσιες μεταφορές να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Ο κύριος Φλέκενστάιν λέει, μίλησε για το υγροποιημένο αέριο ε, και ε, αναφέρθηκε στα 35 χρόνια ε, και εγώ θα αναφερθώ στην πυρηνική τήξη. Εδώ και 40 χρόνια λένε θα γίνουν τα πράγματα τέλεια. Και δεν έγιναν. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να είμαστε επιστημονικά ουδέτεροι. Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί. Αυτό που παίζει ρόλο είναι το αποτέλεσμα. Το πώς θα το πετύχουν δεν έχει καμία σημασία. Αλλά οι τιμές πρέπει να είναι σωστές για να σώσουμε το περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν αυξηθεί το κόστος των θαλασσίων μεταφορών, ε, αυξηθεί το κόστος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε και για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ για την πρότασή σας. Η Επιτροπή παρακαλώ. Κριστιαν Βήμερ uh, uh, ονομάζομαι και δουλεύω στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής για το θείο. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τις τόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα και ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Η συζήτηση μερικές φορές επικεντρώνεται ε, πολύ περιορισμένα στην ναυτιλία. Εγώ θέλω να δούμε κάπως αλλιώς τα πράγματα. Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να έχουμε την ομοθεσία αυτή είναι ο στόχος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσει την ποιότητα του αέρος. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά από τις προδιαγραφές αυτές που θέλουμε να πετύχουμε και γι' αυτό εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα για την ανθρώπινη υγεία εξαιτία δηλαδή της κακής ποιότητας του αέρος. Έχουν γίνει βέβαια από διάφορες χώρες πολλές προσπάθειες με μείωση των εκπομπών, με αφαίρεση 80% τα τελευταία 20 χρόνια του θείου και τώρα για να σας τα πω κάπως πιο σύντομα, τώρα έχουμε φτάσει στην αυτιλία. Τώρα έχοντας ε, καταφέρει στην ξηρά να μειώσουμε τις εκπομπές θείου, τώρα ασχολούμαστε με τη θάλασσα και θέλουμε να μειωθούν και εκεί οι εκπομπές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η ναυτιλία είναι ε, μία σφαιρική επιχείρηση. Μερικές φορές δημιουργούνται από αυτήν προβλήματα, περιφερειακά προβλήματα, αλλά οι λύσεις πρέπει να είναι καθολικές. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη μας τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε για την αυτιλία να προχωρήσουμε συμβάσεις ε, που υπάρχουν για ελεύθερη κυκλοφορία, γιατί είναι αδύνατον ε, μονομερός να εφαρμόσουμε κάτι για χαμηλές εκπομπές. Ε, δουλεύουμε λοιπόν στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και ό,τι διατάξεις υπάρχουν εκεί ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία ώστε να τεθούν στη συνέχεια σε εφαρμογή. Επιπλέον, πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι και να θέλουμε να εφαρμόσουμε πρέπει προηγουμένως να περάσει από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Και η δήλωση για τις περιφερειακές θάλασσες είναι κάτι του οποίο πρέπει να προηγηθεί μια καλή ανάλυση κόστους και κέρδους και να δούμε και τι επιπτώσεις θα έχει στον ανταγωνισμό που δεν μπορούμε να το πούμε τώρα με την απόσταση αυτή των 20 μιλίων. Πάντως, όταν οι κανόνες, το 2015 οι κανόνες του ΠΕΘΑ, το περιεχόν δηλαδή ελέγχου εκπομπών θείου θα αρχίσουν να τεθούν σε εφαρμογή, τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Πάντως, η εισαγωγή νέων προδιαγραφών ποιότητας αποτελεί μία τεχνική πρόκληση για μας. Βλέπω ότι πολλοί, πολλές πλευρές ζητούν επάξη και μια ρήτρα για την προμήθεια θείου. Εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η ρήτρα για την προμήθεια καυσίμων είναι κάτι πιο περίπλοκο, είναι στο παράρτημα 6 και αποτελείται από διάφορα στοιχεία και όχι μόνο από το ελεύθερο πέρασμα, αλλά αναφέρεται επίσης και για τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά αλλά επίσης έχει και μία απέτηση ε, αναφορά σε περίπτωση δηλαδή που κάποιο πλοίο δεν έχει τη σωστή ποιότητα καυσίμων. Πρόκειται για ένα σύνολο δηλαδή και θέλω να σας ενθαρρύνω να δείτε όλες τις πτυχές του κανονισμού αυτού. Οι αλλαγές στον τρόπο μεταφοράς φυσικά είναι ένα μεγάλο θέμα όντως υπάρχει αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Και υπάρχουν δύο τρόποι εδώ για να δούμε το θέμα. Μπορεί κανείς να δει το κόστος για ένα συγκεκριμένο σκάφος, όπου μπορεί τα καύσιμα να αποτελούν το 45% του καθημερινού κόστους ε, λειτουργίας. Από την άλλη μεριά ε, μπορεί όμως κανείς να το δει και διαφορετικά, να δει ε, ποιο είναι το αποτέλεσμα επενδύοντας κάθε ευρώ τι κέρδος έχουμε. Η δικιά μου πρόταση λοιπόν είναι η αξιολόγησή μας να γίνει διαφορετικά, να μην ζητάμε εξαιρέσεις για κάποιες ομάδες, απλώς να λάβουμε υπόψη μας μερικές πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να βρεθούν λύσεις μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο που θέτει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Και κάτι άλλο, για τα τελευταία μέτρα. Όταν δούμε το κόστος εφαρμογής για ολόκληρο τον ε, κλάδο, αυτός είναι χαμηλότερος εφόσον γρήγορα έχουμε νομική βεβαιότητα. Η έλλειψη νομικής βεβαιότητας ανεβάζει το κόστος. Ωραία. Ε, η συγγήτρια για να συνοψίσει παρακαλώ και να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά, ε, για να τελειώσουμε θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τη στήριξή τους, ακόμα και αν υπήρξε διάσταση απόψεων μερικές φορές. Και θέλω να καθησυχάσω αυτούς που ακόμα έχουν τις αμφιβολίες τους. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο και το παράρτημα εγκρίθηκε το 2008. Έχουν περάσει τρία ολόκληρα χρόνια από τότε και έχουμε και άλλα τρία. Κύριε Ήταλα, Ίσως θα μπορούσατε να κοιτάξετε και άλλα θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί ακόμα και αν δεν είχαν υπάρξει κατάλληλες έρευνες. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω εδώ να σας αφήσω την εντύπωση ότι εγώ θα είμαι υπεύθυνη για την εξαφάνιση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Όχι, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Άρα εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο το θέμα της πίστης, ούτε περιμένουμε από κανέναν Άγιο Βασίλη να μας βοηθήσει. Πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι ότι δίποτε άλλο εμένα δεν ε, με καθησυχάζει. Φυσικά, είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το τι θα ακολουθήσει και πώς θα εξελιχθούν οι μεταφορές. Είμαστε όμως εξίσου υπεύθυνοι και για τις πράσινες μεταφορές. Θα θυμόσαστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε την έκθεση Γκρέσ Δεν είναι δυνατόν εγώ να ψηφίζω διαφορετικά τη μια εβδομάδα και διαφορετικά την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τρία χρόνια να καταλήξει στην πρόταση αυτή. Αν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, ίσως να είχαμε μπορέσει να προχωρήσουμε περισσότερο. Ίσως να είχαμε καταφέρει να έχουμε έτοιμη την υποδομή που μας χρειάζεται και τους σταθμούς προμήθειας. Πάντως πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τις επιχειρήσεις. Να ξέρουν ότι δεν θα συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα επιχειρήσεις. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος, και η γνωμοδότηση μετά θα πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου θα ψηφίσουν τον Ιανουάριο. Επόμενο θέμα τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι ο προπολογισμό και, απολογή, και η απαλλαγή. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω το κείμενο, το βλέπετε φαντάζομαι, το έχετε στη διάθεσή σας κι εσείς. Κοιτάξτε, Κάναμε μία διαπίστωση για το τι διακυδεύεται εδώ όσον αφορά τις υποχρώσεις, τις πληρωμές σε σχέση με τις μεταφορές και τον τουρισμό. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα εκείνο το οποίο έχει να κάνει και με το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Γιατί υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα της Επιτροπής μας. Είπαμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο πάλι λαμβάνει υπόψη άλλους τομείς εκτός των μεταφορών και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την σχέση ε, υποχρεώσεων και πληρωμών στην περίπτωση αυτής της συγκεκριμένης απαλλαγής. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια σχετική μείωση όσον αφορά την ε, τήρηση των πληρωμών. Είναι κάπως λιγότερες από ό,τι ήμασταν ε, συνηθισμένοι από 91% ενώ ήταν περισσότερο παλιά. Και αυτό μένα με εξέπληξε, διότι το θέμα με τα δίκτυα είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν στο 100% των πληρωμών για τα δίκτυα εφόσον έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε μπορεί να μας το εξηγήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχομαι τώρα στις άλλες πτυχές που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Παράγραφος 10. Εδώ λέω ότι είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητά μας να παρέμβουμε. Στην περίπτωση του τουρισμού Αυτά τα οποία είπαμε ήταν η αναγνώριση του πώς έχει προετοιμαστεί το θέμα και είπαμε ότι θα έπρεπε η στρατηγική μας να είναι πιο φιλόδοξη ξεκινώντας από την νομική βάση. Εδώ δεν ε, έχει συμπεριληφθεί το τμήμα του προπολογισμού, αλλά θα υπάρξει κάποια τροπολογία για να μιλήσουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παράγραφο 9 Υπάρχει το θέμα της ταχύτητα με την οποία έχουν προχωρήσει προγράμματα όπως ο Γαλιλαίος. Ίσως θα έπρεπε εδώ να αναγνωρίσουμε με κάποια τροπολογία ότι ήδη μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει το θέμα, να το αναγνωρίζουμε αυτό δηλαδή, αν μη τι άλλο. Ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα και άρα μπορεί κάλλιστα να πετύχει. Τέλος, έπρεπε έτσι καλλιώς να περιοριστούμε στο κείμενο, αλλά νομίζω και σας την προτείνω αυτή την τροπολογία, νομίζω ότι θα έπρεπε να προσθέσουμε μια τροπολογία η οποία να αναγνωρίζει τη δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το mid-term review των διευρωπαϊκών δικτύων. Ήταν πολύ επικίνδυνο στην αρχή το χείρημα αυτό γιατί ήταν περισσότερο μια γενική διεύθυνση δαπανών παρά ελέγχου προπολογισμών. Όμως νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον εδώ να αναγνωρίσουμε ότι έγινε τελικά από τη γενική διεύθυνση μου και όχι από κάποια άλλη και ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γενικευθεί και εν ώψη των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών να ζητήσουμε κάτι αντίστοιχο να γίνεται και με άλλα προγράμματα το οποίο να μην είναι καθαρά διευρωπαϊκά δίκτυα, να είναι η έρευνα, για παράδειγμα, η βιομηχανία κλπ. Είναι δηλαδή μια άσκηση πολύ θετική για την απαλλαγή, γιατί έτσι επαληθεύουμε ότι και σε άλλους τομείς για τους οποίους τσακωνόμαστε στο να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση κάθε φορά στις μεταφορές, να απαιτήσουμε την ε, ίδια καλή διαχείριση και να μας το διαβεβαιώνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πάντα μας το ζητάει, αλλά δεν κάνει πάντα την αναθεώρηση αυτή έτσι όπως χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, αν έχετε κάποια άλλη πρόταση, ευχαρίστως να την ακούσω. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι για τα θέματα ασφάλειας μπορεί να υπάρχει εδώ κάποιο έλλειμμα. Ελπίζω στις επόμενες προτάσεις να λυθεί αυτό. Και για τα διάφορα ιστορικά προγράμματα, Μάρκο Πόλο κτλ. υπάρχει και εδώ σημαντική πρόοδο. Ελπίζω λοιπόν πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο, από εκεί και πέρα περιμένω τα σχόλιά σας. να θυμίσω στα μέλη ότι έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω την Αγιάλα Σέντερ για την εξαιρετική της δουλειά. Ερχόμαστε με μια κάποια καθυστέρηση στον προϋπολογισμό του 10 αλλά είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε κάποια σημεία στα οποία εμένει η Επιτροπή στα πλαίσια αυτής της αβέβαιης συγκυρίας και κάτι το οποίο απασχολεί και την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ξέρετε ότι και με την πρωτοβουλία για τα project bonds έχουμε την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό για τη διασύνδεση της Ευρώπης ή στην Ευρώπη, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την Επιτροπή μας να βρει συμπληρωματικές μορφές χρηματοδότησης και από τις ομολογίες της ευρωπαϊκές, τις οποίες βέβαια δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο. Ε, το δίκτυο έχει εξαντλήσει τις πιστώσεις υποχρεώσεων και αυτό αποδεικνύει ότι τα πράγματα προχωρούν. Θα ήθελα εδώ να θυμίσω ότι η μεγάλη σημασία που έχει να έχουμε ισόρροπες οικονομικές συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τις διαμεθοριακές προσπάθειες και προγράμματα. Ένα σημείο είναι το πρόγραμμα Κέσσαρ. Ένα τμήμα των πιστώσεων υποχρεώσεων πήγαν σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού για το 10. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διεκδικούμε ουσιαστικές μειώσεις διοξιδίου του άνθρακα από τις αερομεταφορές και από την άλλη να μειώνουμε ταυτόχρονα το Κέσσαρ. Είναι λίγο δύσκολο τώρα για τον τουρισμό πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου έτσι ώστε να συνεχίσουμε την καλή πρακτική που έχουμε πετύχει σε διάφορες περιοχές ε, άλλες. Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και βέβαια να ρυθμίσουμε κάποιες διοικητικές διαδικασίες που αμφισβητούν, αν θέλετε, την επιτυχία της προσπάθειας την οποία εμείς κάνουμε. Κύριε Μάιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για όλα αυτά που μας προτείνει. Ε, συμφωνώ απόλυτα. Ε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Καταρχήν το σημείο υπερθυμών 3 αναφέρεται ότι το ποσοστό απορρόφησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι πολύ ψηλό και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μου αρέσει επίσης το ότι η συγγήτρια αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν κάτι έτσι ώστε να βελτιωθεί ε, περαιτέρω η χρηματοδότηση σε αυτόν τον σημαντικό τομέα των ε, υποδομών. Όσον αφορά τώρα την προοπτική του μέλλοντος, ε, χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ε, και τα περίφημα ομόλογα χρηματοδότησης έργων, αναφέρουμε στο σημείο υπαριθμών 5, ε, πράγματι πρέπει να χρηματοδοτηθούν πλέον αυτά τα ομόλογα. Έχω μια παρατήρηση, νομίζω στο γερμανικό τουλάχιστον κειμενό λείπουν τρία μηδενικά. Γίνεται λόγος για, τρία, με για 10 εκατομμύρια, είναι 10 δι Ξέρουμε πολύ καλά βέβαια όλοι μας τα ποσά. Εντάξει, δεν πειράζει που λείπουν τα τρία μηντονικά. Εγώ απλά το είπα για να το διορθώσετε. Και κάτι άλλο ε, για τον τουρισμό. Ε, τώρα πλέον έχουμε νέες αρμοδιότητες και ε, δεν προβλέπονται ακόμα τα κονδύλια που θα επιθυμούσαμε έτσι ώστε να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Είναι όμως θετικό το γεγονός ότι η συγκήτρια καλεί την Κομισιόν ε, να καταθέσει πολιτή προγράμματα. Σε γενικές λοιπόν γραμμές, πολύ καλή δουλειά και εμείς τη δεχόμαστε και συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Αγιάλα Σενδέρ. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, παράγραφος 2. Αναφερόμεθα στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις στρατηγικές μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει πιο συνεκτικά τα προγράμματα συνοχής με τα προγράμματα που ε, έχουν σχέση με την Ατζέντα 2020 και με τις ελλείψεις στον τομέα της ενέργειας σε σχέση με τις ανάφορες. Ε, δεν δίνουμε προσοχή σε σχέση με τη διαχείριση της ζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου ε, με την ζήτηση. Ασχολείται μόνο με την προσφορά. Στην παράγραφο 3 θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης την πράσινη βίβλο του Απριλίου 2009 που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ένα κατάλογο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού από τα διαφορετικά ταμεία από τη μία και από άλλες πηγές από την άλλη. Τρίτον, να αναφερθώ στα Connecting Europe Facilities. Ίσως είναι λίγο πρόωρο αυτό γιατί η τελική απόφαση δεν έχει πλέον, δεν έχει ακόμα ληφθεί. Και μια τελική παρατήρηση για το Κέσαρ. Θα ήθελα κάποιες εξηγήσει, περισσότερες εξηγήσει, γιατί οι δαπάνες ε, υπερέβησαν τις προβλέψεις. Ελπίζω και τα αποτελέσματα να υπερέβησαν τις, ε, ε, τα, αποτελέσματα να ήταν περισσότερα από όσα εν πάση περιπτώσει περιμέναμε. Γιατί δεν νομίζω τελικά ότι έχουμε μειώσει όσο θα θέλαμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις αερομεταφορές. Δώστε μας λοιπόν εξηγήσεις κύριος Μπελούτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω τον τουρισμό, διότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Κατά τα άλλα θα ήθελα να πω ε, The review made into... Το TNT έχει προχωρήσει αρκετά καλά. Ήδη το 2011 ξεκινήσαμε μια νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος και πέρα από την επιβράδυνση που έχει προκληθεί από την οικονομική ύφεση, η δημοσιονομική πρίκα θα έλεγα των προγραμμάτων αυτών είναι σχετικά ικανοποιητική. Έχουμε βελτιώσει τις προβλέψεις για όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες Μπορείτε να δείτε αυτό και στην ικανοποίηση την οποία εξέφρασε και το ελεγκτικό συνέδριο. Μία παρατήρηση για τον Μάρκο Πόλο. Το 2009 είδαμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. έγιναν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, μικρορυθμίσεις και κάποιες από τις πιστώσεις χρηματοδότησαν άλλα προγράμματα, όπως είχατε προτείνει και εσείς. Κατά τα άλλα, οι άλλες εξωτερικές υπηρεσίες λειτουργούν καλά, έχουν καλές επιδόσεις. Μία μικρή μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, η οποία είναι φυσιολογική θα έλεγα γιατί όταν δεν παίρνει κανείς τις αποδείξεις δεν μπορεί να ε, πληρώσει. Ε, γενικά ο, κανο, ο, τομέας μας είναι ικανοποιητικά λειτουργικός, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κυρία Γιάλα Σενδέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ή εγώ δεν το έχω βρει εδώ ή δεν το κατάλαβα στην απάντησή σας, αλλά εγώ κάτι σας ρώτησα. Σας ρώτησα για την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές φέτος ιδιαίτερα, ε, για τον προπλωσμό δηλαδή 2010 στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Διότι η σύγκριση δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί μειώθηκε, αν είναι αυτό που είπατε. Τώρα για τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι και που βρίσκω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα για το Σέζαρ. Ναι, ευχαρίστως να βρω τροπολογίες σας προκειμένου να δείξουμε τι θέλουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισμό. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε εδώ τα σχόλιά μας με τροπολογίες. Στην κυρία Ντυρόν θέλω να πω ότι δεν ξέρω αυτή η γαλλική μετάφραση, αλλά στο σημείο 4 πολύ συγκεκριμένα μιλάμε για το Connecting Europe, για το μηχανισμό δηλαδή για τη διασύνδεση στην Ευρώπη, που είναι τα VEDM. Εγώ ήθελα ακριβώ να υπάρχει. Και παρά τον κανονισμό που υιοθετήθηκε πρόσφατα, μπορούμε εδώ να πούμε ότι μας ενδιαφέρει. Αυτά. Και μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Δεν λέω ότι είναι πρόβλημα, αλλά είναι ένα περίεργο στοιχείο και θα ήθελα να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μπανούτσι, μήπως θα μπορούσατε να μας απαντήσετε σύντομα από αυτού. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το Caesar και μετά θα πάω στα TNT. Όπως ξέρετε, το Σίζαρ έχει χάσει την ε, ταχύτητά του. Γι' αυτό κάποιες ε, πληρωμές έχουν καθυστερήσει τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον. Τώρα αποκτά εκ νέου ε, την ταχύτητά του και απορροφά τα όσα είχαν μείνει την προηγούμενη περίοδο. Απορροφάει τα κονδύλια δηλαδή πιο γρήγορα. Τώρα για το θέμα των τεντή Το κύριο πρόγραμμα είναι ένα πολιετές πρόγραμμα. Αυτό το οποίο έγινε στα τέλη του 2010 ήταν αναθεώρηση των προγραμμάτων τα οποία είχαν μείνει πίσω, είχαν καθυστερήσει. ή τα ποσά για τις πληρωμές, που δεν έχει αυτό καμιά σχέση με τις υποχρεώσεις, χρησιμοποιήθηκαν για να ξαναγίνουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος, ναι διαγωνισμοί δηλαδή. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τα προβλεπόμενα κονδύλια για ολόκληρη την περίοδο. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο, κύριε Βανουτζή. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι στι 12 το μεσημέρι στι 11 Ιανουαρίου. Θα ψηφίσουμε εδώ το Φεβρουάριο. Μετά η συνταγματική, η διορθώνει ο Πρόεδρος, η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού θα ψηφίσει τον Μάρτιο και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Μάιο. Λοιπόν, η πρώτη ημερομηνία που σας έδωσε ήταν 11 Ιανουαρίου, ψηφίσουμε εδώ. Επόμενο θέμα είναι η απαλλαγή για τους οργανισμούς και το ΣΥΖΑΡΟ. Κύριε κύριος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, είδαμε αυτές, αυτούς τους τέσσερις οργανισμούς και συνολικά στην πρόταση μου ως ε, κατατίθεται ε, προτείνουμε την απαλλαγή στην ΕΜΖΑ εκεί αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι η ΕΜΖΑ τηρεί κατά γράμμα αυτά που τους είπε πέρυσι το ελεγκτικό συνέδριο τις παρατηρήσεις του. Κυρίως ότι όσον αφορά τις προσλήψεις έπρεπε να αλλάξουν τη διαδικασία και την άλλαξαν. Όσον αφορά τον Οργανισμό για την Ενέργεια Ασφάλεια, και εκεί υπάρχουν ε, επικριτικές παρατηρήσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σχετικό, προτείνεται η απαλλαγή. Όσον αφορά ε, τον οργανισμό ΣΕΖΑΡ, εκεί πρέπει να επισημάνουμε ότι δύο γραμμές του προεπολογισμού, δηλαδή τα διοικητικά έξοδα και η γραμμή για τις μελέτες, ε, ξεπεράστηκαν αυτές τις γραμμές ε, κατά 10 ή 11, αντίστοιχα 11%. Αυτό δεν μπορεί να είναι μόνιμη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως ε, προτείνουμε ο, ο διευθυντής αυτών των οργανισμών οι διευθυντές να λάβουν απαλλαγή. Και στους ευρωπαϊκούς σιδηρόδρομους έχουμε ένα πρόβλημα που έρχεται και επανέρχεται. Αυτή τη φορά μιλάμε για 5,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Ε, ε, και πέρυσι το είπαμε αυτό, ότι και αυτό δεν μπορεί να είναι μόνιμη κατάσταση. Βέβαια, του χρόνου, αν έχω καταλάβει καλά, ε, θα έχουμε να συζητήσουμε για αναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών. Τότε λοιπόν θα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να συζητήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Πάντως και στον οργανισμό αυτό, ε, τον οργανισμό των ε, σιδηροδρόμων και σε αυτόν επιθυμούμε να χορηγήσουμε απαλλαγή. Έτσι λοιπόν ε, και στις τέσσερις περιπτώσεις λέμε ναι, απαλλαγή, συμφωνούμε, σηκώνουμε θετικά το χέρι, έστω και αν τρέμει λιγάκι λέει χαρακτηριστικά ο μιλητή. Κυρία Μπλάστο. Το ΖΕΖΑΡ, όπως είπατε, εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο πλέον. Και συμφωνώ με τον κύριο Φλέκενστάιν σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2010. Παρ' όλα αυτά, έχω κάποιες μικρές επιφυλάξεις για την διαχείριση ιδιαίτερα του σιδηροδρομικού κομματιού. Η Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Υπηρεσία θα πρέπει να σεβαστεί, θα έλεγα, τον ετήσιο χαρακτήρα του προϋπολογισμού. Δεν είναι φυσιολογικό να αναβάλλεται από τη μία χρονιά το πρόγραμμα για την επομένη και να μεταφέρονται τα χρήματα που έχει στη διάθεσή της από τη μία χρονιά στην άλλη λόγω ακριβώς των προβλημάτων στις αγορές. <clears throat> Είναι επίσης σημαντικό να ολοκληρώσουμε ταχύτατα την αναπτυξιακή πρώτη φάση του ΖΕΖΑ. Αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα να μειώσουμε τις εκπομπές καυσαερίων, να καταστήσουμε ρευστές τις μεταφορές και να θα έλεγα πρασινίσουμε τον ευρωπαϊκό αεροπορικό χώρο. Γι' αυτό λοιπόν το Σέζαρ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει <clears throat> ότι περίσευμα υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 57 εκατομμύρια ευρώ. Ανησυχώ και για τις κριτικές οι οποίες διατυπώθησαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφάλειας ε, στις, ε, στους διαγωνισμούς τους οποίους οργανώνει. Αλλά είπατε ότι αυτά θα τα πούμε το Φλεβάρι βέβαια. Πάντως δεν είναι ε, δυνατόν να ανεχθούμε προτιμησιακές συμπεριφορές και διακρίσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου να πιέσει επιτέλους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει με τη σειρά της εξηγήσει από την ΑΕΣΑ, η οποία υπενθυμίζω υφίσταται σε εισαγωγικά τους κοινοτικούς κανόνες και ρυθμίσεις για τους διαγωνισμούς κτλ. Δεν θα πω τίποτα για τις θαλάσσιες μεταφορές. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έκανε παρατηρήσεις γύρω από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις θαλάσσιες μεταφορές. Μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Κνούτ Φλέκενστάιν. Πράγματι γνωρίζουμε ότι οι οργανισμοί αυτοί σε γενικές γραμμές προσφέρουν καλή δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε και κατά την κατάρτιση του προπλογισμού ότι δεν πρέπει να λάβουν περισσότερα κονδύλια αλλά να παραμείνουν ε, σε αυτά που έχουν εκτός από την έμψα. Αυτό το εγκρίναμε στην τελευταία ολομέλεια. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Φλακνιστάν και στην αλληλουχία. Η έμψα είχε κάποιες μαύρες κοιλίδες, εξαφανίστηκαν αυτές ε, και η έμψα ήταν η καλύτερη. Στην Ιάσα, αυτό το είπε και η κυρία Βλάστο μόλις τώρα, το θέμα είναι πώς λειτουργούν οι διαγωνισμοί και πώς γίνεται η επιλογή του προσωπικού. Αυτό όμω δεν είναι και τόσο τραγικό, έτσι ώστε να πει κανείς, α, γι' αυτό δεν τους χορηγούμε απαλλαγή. Όσον αφορά ε, στην ΣΕΖΑΡ, την κοινή επιχείρηση ΣΕΖΑΡ, νομίζω ε, πρέπει να δούμε λιγάκι τις διοικητικές δαπάνες ε, που ξεπερνιόνται κατά 11 περίπου 100. Αυτό είναι πάρα πολύ. Στις μελέτε και τις έρευνε. εντάξει, είναι σημαντικέ οι μελέτε, αλλά οι διοικητικέ δαπάνε που αυξάνονται τόσο πολύ ε, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να τους ε, ε, εκφράσουμε, να τους αποδώσουμε μομφή για τους σιδηρόδρομους. Δεν είμαι και πολύ σύμφωνη, αλλά τέλος πάντων ας τους δώσουμε απαλλαγή, γιατί και πέρυσι τους κάναμε την διαπροειδοποίηση ότι μεταφέρουν και πάλι ποσά. Η μομφή δεν αρκεί νομίζω. Εντάξει, ας τους δώσουμε απαλλαγή, αλλά παρόλα αυτά παραμένει πρόβλημα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Και διαρωτώ με κατά πόσον θα το πράξουν αυτό. Αν εκφράζουμε απλώς μια αιμομφή, δεν ξέρω αν την παίρνουν σοβαρά υπόψη. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάτι πιο αυστηρό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα καταθέσω τροπολογία με αυστηρότερο ύφο, ε, γιατί δεν είναι δυνατόν να κάνουν συνέχεια τα ίδια και δεν πρέπει του χρόνου να επαναληφθούν τα ίδια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Ντουρά. Για το Ζέζαρ θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Βλάστο για την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των αερομεταφορών, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς το 11% αύξησης των διοικητικών δαπανών θα επιταχύνει τη διαδικασία για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Το θέμα αυτό των ενιαίων ευρωπαϊκών ουρανών είναι πολιτικό θέμα και εδώ δεν θέλει το Συμβούλιο να προχωρήσει. Οπότε πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε τη σύνδεση ανάμεσα στο ΖΕΖΑΡ και τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτό είναι θέμα πολιτικό και πρέπει να επιληθεί σε επίπεδο συμβουλίου. Και το ΖΕΖΑΡ θα πρέπει να μας εξηγήσει το 11% αύξηση των διοικητικών δαπανών. Δεν θα πρέπει για το ΖΕΖΑΡ να πέσουμε στο ίδιο σενάριο με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία επιθυμούμε ή όχι, αλλά τα οποία πάρα πολύ συχνά αυξάνουν τις δαπάνες τους με πολύ μεγάλο ρυθμό και με ανεξέλεγκτο θα έλεγα πολλές φορές ρυθμό. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε κόκκινη κάρτα για το ΖΕΖΑΡ. Είναι πολιτικό το πρόβλημα και δεν θα πείσει το ΖΕΖΑΡ τα κράτη-μέλη σχετικά με τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς, δυστυχώς. Ρίκε. Ευχαριστώ. Μία πρώτη γενική παρατήρηση για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι κοινοτικά μέσα οι εξωτερικές υπηρεσίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επιμένει σε σχέση με τα θέματα αυτά πρέπει να φροντίζει τις υπηρεσίες αυτές. Αλλά επειδή τους αγαπάμε πρέπει να τους ζητήσουμε να είναι καλοί. Λοιπόν, τώρα για το σιδηροδρομικό πακέτο. Υπάρχουν συγκεκριμένες καθυστερήσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες εδώ και τρία χρόνια. Να πούμε ότι είναι η τελευταία βέβαια υπηρεσία αυτή για το σιδηρόδρομο, η οποία τέθηκε σε λειτουργία. Έχει δυσκολίες και την επιφορτίζουμε με αποστολές οι οποίες δεν είναι στα μέτρα της αν θέλετε. Δύο παραδείγματα. Όταν του ζητάμε ε, γνωμοδοτήσεις για διαφορές ανάμεσα σε εμπλεκόμενους, ας πούμε. Όταν του ζητάμε να κάνει εκθέσεις για σιωδρομικά ατυχήματα, σαν και αυτό που είχε γίνει πριν 1,5 χρόνο. Ε, πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε. Ή από τη μία δεχόμαστε ότι του ζητάμε να λειτουργήσει ε, <clears throat> κατά από συνθήκες, δεύτερον να βρει το σωστό προσωπικό τρίτον να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει και τέταρτον να μας δίδει και εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης όπως ε, όταν τις χρειαζόμαστε συνεπώς. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αρμοδιότητες και τον κανονισμό της υπηρεσίας για τους αεροδρόμους. Δεν μπορούμε να αντιζητάμε τα πάντα πάντα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα βελτιωθούν τα πράγματα. Καλό είναι να λέμε ότι οι καθυστερήσεις δεν είναι επιθυμητές, από την άλλη δεν θα πρέπει και να τις προκαλούμε. Και Μπονούτσι για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. Για το αέρα. είναι μια κατάσταση την οποία γνωρίζουμε εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια. Η υπηρεσία αυτή πράγματι είναι σχετικά αργή σε επίπεδο διαγωνισμών. Έχουν φτάσει στο τέλος του χρόνου και θα πρέπει να εκτελέσουν τις αποφάσεις που πήραν τον επόμενο χρόνο. Αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε και δημοσιονομικές μεταφορές αρκετά υψηλές. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι και άλλες μέθοδοι, να χρησιμοποιήσουν άλλες μεθόδους όπως, όπως ε, τα προγράμματα πλαίσιο για να επιταχύνουν τις καταστάσεις αυτές στο μέλλον, να τα επιταχύνουν τη λειτουργία τους καλύτερα στο μέλλον. Για το Σέζαρ θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους από το Σέζαρ γιατί νομίζω ότι έχουμε μια σύγχυση ανάμεσα στις διοικητικές δαπάνες για το Σέζαρ με άλλου είδους δαπάνες. Οι διοικητικέ δαπάνες για το ΖΕΣΑΡ παραμένουν πάντα στο ανώτατο όριο. Λέγομαι Μποργκίνη από το ΖΕΣΑΡ. Όπως είπε ο κ. Μπονούτσι, οι διοικητικέ δαπάνες για το ΖΕΖΑΡ παραμένουν στις πιστώσεις υποχρεώσεων που είχαν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχει περάσει δηλαδή το όριο. Η παρατήρηση του ελεγκτικού συνεδρίου λέγει ότι σε επίπεδο πιστώσεως υποχρεώσεων το επίπεδο εκτέλεσης ξεπεράστηκε κατά 11% και κατά 9% στις δύο γραμμές του προϋπολογισμού και αυτό καλύφθηκε από πιστώσεις πληρωμών οι οποίες ήταν διαθέσιμες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε ξεπεράσει λοιπόν τις διοικητικές μας δαπάνες, τον προϋπολογισμό που είχαμε. Ευχαριστώ. Φλέκενστάιν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. ο κύριος Μπελούτσι θέλει να επανέλθει για την υπηρεσία για τις, για τις αερομεταφορές. Να σας πω ότι άλλαξε το λογιστικό στη σύστημα το 2010 η ΕΑΖΑ για να το εξυγχρονίσει και να ταυτιστεί με αυτά τα οποία γίνονται και στις άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Αυτό θα λύσει εν μέρη το πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε ήταν οι προσλήψεις για την ΕΑΖΑ. Άλλαξαν και εκεί τις διαδικασίες που ακολουθούσαν και νομίζω ότι καλύπτεστε τώρα. Δεν νομίζω θα δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ ο κύριος Φλέκενστάιν. Ακόμα καλύτερα αν τα πράγματα πάνε καλύτερα στην ΕΑΖΑ. Απλά χρειάστηκαν κάποιο χρόνο μέχρι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ε, την επίπληξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Να πω μόνο κάτι για την αίρα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση ε, η επίπληξή μας να είναι πιο αυστηρή. Εγώ δεν θέλω να αρνηθώ την απαλλαγή, αλλά μπορούμε να καταστήσουμε σαφές ότι αν αυτά επαναληφθούν την επόμενη χρονιά, τότε δεν θα ξαναδώσουμε ε, απαλλαγή γιατί είμαστε δυσαρεστημένοι. Πολύ ωραία. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για αυτήν την έκθεση είναι 11 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Ε, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών το Φεβρουάριο και μετά θα υπάρξει η ψηφοφορία στον Ολομέλεια το Μάιο. Όπως λοιπόν και με άλλες ε, τις εκθέσεις περί απαλλαγής, ε, η ε, προθεσμία είναι 11 Ιανουαρίου. Το επόμενο θέμα είναι τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Τέιλορ, που εξαφανίστηκε όμως, που είναι καθοδόν. που σημαίνει να πω εγώ μερικά πράγματα. Θα θυμάστε ότι είναι δική μας αίτηση πρωτοβουλίες ε, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα ε, των ε, δικαιωμάτων των επιβατών στην περίπτωση που υπάρχει άρνηση επιβίβασης ή ακύρωσης της πτήσης και γίνεται λόγος και για την κινητικότητα των επιβατών που έχουν προβλήματα κινητικότητας. Ελπίζω ο κύριος Τέιλορ θα ε, κοινοποιήσει τις απόψεις του. Ο κύριος, κύριε Τέιλορ, ήρθε ο κύριος Τέιλορ, ε, θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Δεν ξέρω, είναι παρούσα και η Κοινωνική Επιτροπή. Ας εξετάσουμε πρώτα την έκθεση του κυρίου Τέιλορ.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 Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους και ε, να ευχαριστήσω τις ΜΚΟ και τις ε, ειδικέ οργανώσεις που βοήθησαν, να ευχαριστήσω και την Κομισιόν και τους ε, συμβούλους της ομάδας που όλοι αυτοί βοήθησαν να φτάσει η έκθεση στη φάση που είναι τώρα. Στην τελευταία συνάντηση των σκιωδών είχα την χαρά να διαπιστώσω ευρεία συμφωνία στα περισσότερα θέματα. Αυτή λοιπόν έχει ως στόχο να εξετάσει την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού 261 του 2004 και εκεί προβλέπονται κοινοί κανόνες για την αποζημίωση και για την παροχή βοήθειας επιβάτος στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή μεγάλης καθυστέρησης. Επίσης υπάρχει έκθεση Κομισιών για την λειτουργία του κανονισμού 1107 που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και με αναπηρία ή με αναπηρία όταν τα άτομα αυτά ταξιδεύουν. Τα δικαιώματα των επιβατών έχουν τεθεί σε πάρα πολλές, ε, πολλούς κανόνες και νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ κοιτάζω το θέμα από ευρύτερη οπτική γωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ολόκληρη την έκθεση υπογραμμίζω την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, καλύτερη ερμηνεία, να εφαρμόζονται νέα οι κανονισμοί σε ολόκληρη, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι απαραίτητο οι δικαστικές αποφάσεις, η νομολογία ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να συμπεριληφθεί στην ε, επικείμενη στον επικείμενο κανονισμό 261. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η λογοδοσία και η διαφάνεια να ενισχυθούν τα υπάρχοντα δικαιώματα και να είμαστε σίγουροι ότι αυτά είναι απόλυτα σαφή στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η έκθεση αυτή κατατίθεται έγκαιρα επειδή του χρόνου πρόκειται να τροποποιηθεί από την Κομισιόν ο 261 του 2004. Ελπίζουμε λοιπόν όλοι μας ότι ε, θα υπάρξει αναθεώρηση και άλλων νομοθετημάτων όπως ε, η οδηγία για τα αεροπορικά και ειστήριο πακέτο. Ας πάμε τώρα σε αυτή την ίδια την έκθεση. Ε, συνοπτικά θα αναφέρω τα βασικότερα σημεία. Στο ευρύτερο πλαίσιο θεωρώ ότι οι επιβάτες πρέπει να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, να μπορούν να τα διεκδικήσουν, έχουν, να έχουν προσπέλαση στην ενημέρωση. Η ενημέρωση να γίνεται με απλό, εύληπτο, κατανοητό τρόπο ε, σε όλες τις φάσεις του ταξιδιού. Από την ώρα που ο επιβάτης ε, αρχίζει να σκέφτεται κατά πόσο επιθυμεί να αγοράσει ε, εισιτήριο ή όχι. Για να Διασφαλίζονται λοιπόν όλα τα δικαιώματα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Λέω ότι οι αεροπορικέ εταιρείε θα πρέπει σε κάθε ε, αεροδρόμιο που χρησιμοποιούν να έχουν και έναν ειδικό υπάλληλο ο οποίο θα ενημερώνει, θα προσφέρει βοήθεια, θα δίνει την αποζημίωση ή θα ε, βάζει του επιβάτες σε άλλες πτήσει, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην πτήση που έχουν ε, κλείσει, που έχουν κρατήσει να υπάρχουν λοιπόν ειδικοί φορείς ανεξάρτητοι οι οποίοι θα ασχολούνται με τις ε, καταγγελίες ε, των επιβατών, θα βοηθούν στην επίλυση των διαφορών ε, και αν χρειάζεται θα επιβάλλουν και κυρώσεις. Επίσης ζητώ να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών επιβολής κυρώσεων θα συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί μάλιστα ο οργανισμός αυτός ή το δίκτυο θα δημοσιεύει και τα παράπονα, τις καταγγελίες που λαμβάνει. Επίσης αναφέρω ότι οι ανάγκες των επιβατών θα πρέπει να καλύπτουν σε περίπτωση ε, πληρωμών ή πτώχευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Να υπάρχει σωστή εφαρμογή του κανονισμού πλήρης ε, διάβγεια και διαφάνεια τιμών. Αυτό ισχύει και στις ε, καταχωρήσεις και διαφημίσεις ε, των αεροπορικών εταιριών. Οι επιβάτες επίσης πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που δίνουν οι αεροπορικές εταιρείε με βάση το APNR. Οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τις λεπτομέρειες στα εισιτηριά τους στην περίπτωση ε, που έχουν κάνει κάποιο λάθος στην κράτηση. Πόσες φορέ έχουμε ακούσει ότι κάποιος ε, ε, είπε λάθο το όνομά του και όταν ζήτησε να το διορθώσει του ζήτησαν 40 λίρε ή 40 ευρώ για να κάνει μια μικρή διόρθωση στο όνομα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πολύ βασικό δικαίωμα των επιβατών είναι στην, στο ασφαλές ταξίδι. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο όλοι οι επιβάτες, ακόμα και παιδιά κάτω της ηλικίας των 2 ετών, των ετών να έχουν ασφαλή θέση στο αεροπλάνο. Και τέλος, οι επιβάτες ε, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ταξιδιού τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, καλείται η Επιτροπή και οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν τη δουλειά τους που θα επιτρέψουν να υπάρχουν αντικειμενικές συγκρίσεις του περιβαλλοντικού αποτυπώματος διαφόρων αεροπορικών εταιριών και διαφόρων μέσων μεταφοράς. Ε, ο κανονισμός 261 προβλέπει κανόνες για την αποζημίωση, ε, προβλέπει την παροχή βοήθεια στους επιβάτες σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης, μεγάλης καθυστέρησης ή άρνησης επιβίβασης. Ε, η ε, ευκρίνεια, η σαφήνεια είναι το κλειδί. Γι' αυτό λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού 261 ε, να την ενσωματώσει στον νέο κανονισμό, να συμπεριλάβει και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για διάφορους ορισμούς συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών συνθήκων, όπως επίσης και των κανόνων για την αποζημίωση. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να παίξει αυτό το ρόλο μου ζήτησαν ε, να λάβω υπόψη μου ε, να καταρτήσω εγώ έναν κατάλογο αυτών των ε, έκτακτων περιπτώσεων. Αλλά είμαι σίγουρος ότι στον κατάλογο αυτό είναι πολύ πιθανό να μην περιλάβει κανείς κάποια περίπτωση που θεωρεί ιδιαίτερη, αλλά αν συμβεί κάτι και επειδή δεν περιλαμβάνει τον κατάλογο δεν σημαίνει ότι δεν είναι έκτακτη και ιδιαίτερη περίπτωση. Επίσης, αν υπάρξει καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης, πρέπει να ενημερώνεται ο επιβάτης. Η ακυρωση πρεπει να ενημερωνεται ο επιβατης η διαρκεια της καθυστέρησης είναι σημαντική να του προσφερθούν, παραδείγματο χάρη, εναλλακτικέ λύσεις, αλλά και από άλλα μέσα μεταφοράς, αν αυτό είναι δυνατό. Ο, ε, επιβάτης πρέπει να έχει δυνατότητα επιλογή σε τρία πράγματα ε, και αυτό είναι ένα βασικό του δικαίωμα. Επίσης, ε, οι επιβάτες που είχαν την ατυχία οι αποσκευές τους να μην έρθουν ε, να πάνε κάπου αλλού, αυτοί έχουν ε, τα ίδια δικαιώματα σαν ε, να πρόκειται για τους ίδιους, αν και πρόκειται για τις επισκευές. Για να μπορούν οι αεροπορικές εταιρείε να εξετάζουν τις πιο ευάλωτες ομάδες ή επιβάτες πρέπει να μπορούν μόνοι τους να αγοράζουν τα αυτά που χρειάζονται και να ζητούν τα χρήματα από τις αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, ε, η αποζημίωση, τα κριτήρια και οι μηχανισμοί. Αυτά ε, θα πρέπει να αναθεωρούνται από την Κομισιόν υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποδυναμώνονται τα ισχύοντα. Θα ήθελα τώρα να φερτώ λιγάκι στον κανονισμό 1107 που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Πιστεύουμε ότι η ανεμπόδιστη πρόσβαση είναι καθοριστικό στοιχείο για να ε, διασφαλιστεί ισότητα πρόσβασης ε, και για αυτή την ιδιαίτερη ομάδα. Η έλλειψη κατάρτισης του προσωπικού και η φυσική υποδομή των αερολιμένων και των αεροσκαφών αποτελούν εμπόδια που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά διασφαλίζοντας ε, την πρόσβαση ε, στο αεροσκάφος ε, και στις πόρτες του αεροσκάφους να είναι κατάλληλες οι πόρτες για να μπορεί το αμαξίδιο ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο είναι απαραίτητο να φτάσει μέχρι το αεροσκάφος. Είναι επίσης σημαντικό τα πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα και τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να συνοδεύονται εφόσον απαραίτητο από αναγνωρισμένο οδηγό ή βοηθό σκύλο στο αεροσκάφος και να διασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβασή του σε οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς. Τέλος, οποιαδήποτε ζημία στον εξοπλισμό κινητικότητας προσώπων με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να αποζημιώνεται πλήρως εδώ ε, μιλάμε για μια αύξηση από το όριο των 1.200 ευρώ που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ζωτική σημασία για τον ενδιαφερόμενο και είναι και πολύ ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καλύπτεται. Τέλος, η ενημέρωση των προσώπων με μειωμένη κινητικότητα και των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να είναι απολύτως προσιτές και με μορφή που να αντιστοιχεί στις ανάγκες τους. Αυτά είχα να πω εν είδη εισαγωγή ε, κύριε Πρόεδρε και με μεγάλη μου χαρά περιμένω να ακούσω τι έχουν να πούν οι σκιώδεις ηγητές και βεβαίω η Επιτροπή. Uh, ο κύριος Νάντες Βαταγιά είναι εδώ από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που είναι η συγητής της Επιτροπής εκείνης οπότε για το ίδιο αυτό θέμα, ε, οπότε παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέσω των τμήματων της που ασχολούνται για τις μεταφορές ε, έλαβε την επιστολή του Προέδρου σας με ερωτήσεις σχετικά με τους δύο αυτούς κανονισμούς, τον 261 και τον 1107. Εμείς δύο φορές συνεδριάσαμε και είχαμε και μια δημόσια ακρόαση, μάλιστα με τους ενδιαφερόμενους τομείς, κλάδους. Καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα που θα σας μεταφέρω κάπως συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα, όλοι όσοι συμμετείχαν στην ακρόαση πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση. Και αυτό γιατί οι δύο κανονισμοί, κυρίως ο 261, δεν είναι αρκετά σαφείς και έτσι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγκάστηκε πολλές φορές να αποφανθεί και να δημιουργήσει νομολογία. Αυτή την νομολογία λοιπόν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τώρα πρέπει να την ενσωματώσουμε σε ένα νέο κανονισμό. Έπειτα πρέπει να δούμε ποιο είναι το εύρος ε, της, ε, και ποια ακριβώ είναι αυτή η έννοια που την ονομάζουμε έκτακτες περιστάσεις. Αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί. Πρέπει να οριστεί δηλαδή καλύτερα αυτή η έννοια των έκτακτων περιστάσεων, για να μην επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες. Και τρίτον, υπάρχει και κάτι άλλο πολύ βασικό, που είναι η αρρωγή προς τον ε, επιβάτη. Εδώ πρέπει επίσης να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή σε τι συνίσταται αυτή η αρρωγή ιδιαίτερα στις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, στην περίπτωση ακύρωσης πτήσεως ή στην περίπτωση καθυστέρησης. Είναι αυτά τα τρία ζητήματα που απασχόλησαν περισσότερο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και εκεί έχουμε επιμείνει περισσότερο σε σχέση με την αρχή. Εμείς εκπονήσαμε μία έκθεση όπου εντοπίζονται τα διάφορα σημεία που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά. Είναι συγκεκριμένα πράγματα όπως η ρύθμιση καταστάσεων που δημιουργούνται στην περίπτωση επαναπρογραμματισμού των πτήσεων, προβλήματα που έχουν να κάνουν να μαχάσει κανείς ε, την επόμενη πτήση που πρέπει να πάρει, τέτοια πράγματα τα οποία αναφέρονται στην εκθεσή μας και φαντάζομαι ότι η γραμματεία σας το έχει δώσει το έγγραφο αυτό. Τέλος, Πρόεδρε, υπάρχει και το θέμα του κανονισμού 1107. Είναι ένας πολύ πρόσφατος κανονισμός αυτός, όμως οι διάφορες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία δεν είναι ικανοποιημένες με την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, έτσι όπως έχει σήμερα. Πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος ή να καλυφθεί με κάποιο ερμηνευτικό σημείωμα για να καλύψει τις περιπτώσεις ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Αλλιώς, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, λένε ότι πολύ συγκεκριμένα θα ζητήσουν την αναθεώρηση του κανονισμού. Έτσι λοιπόν, συνοπτικά, αυτό είναι το περιεχόμενο της δικιάς μας έκθεσης που είναι στη διάθεσή σας εφόσον θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαταγιά που ήρθατε και που μας παρουσιάσατε την ε, έκθεσή σας από την ΟΚΕ. Ο κύριος Σαζάντα, τώρα από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. θα ήθελα... Ευχαριστήσω τον κύριο Τέιλορ για την προσπάθεια την οποία έκανε και θα συμφωνήσω με το μεγαλύτερο κομμάτι των παρατήρησεών του. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες πάντως, οι οποίες θα πρέπει να καταστούν, θα έλεγα, πιο συγκεκριμένες και να γίνουν πιο κατανοητές. Γενικά, είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει ανάγκη να αναδιατυπωθεί ο 261-2004 γιατί τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να περιστιαστούν σε ένα έγγραφο με εμπεριστατωμένο τρόπο. Συμφωνώ με τον εισηγητή επίσης ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αποφασίσουμε ε, το τι εννοούμε έκτακτες συνθήκες. Τρίτον, ακόμα και οι καλύτερες ρυθμίσεις νομικά δεν είναι χρήσιμες αν οι επιβάτες δεν τις γνωρίζουν. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε ενημέρωση σε επίπεδο κοινοτήτων, συγκεντρώνοντας την προσοχή μας από τη μία στη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων των επιβατών από τους ίδιους τους επιβάτες και ταυτόχρονα να ενημερώσουμε τους επιβάτες πώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο. Για το άρθρο 13 του 261-2004 Διευκρινίζεται ότι μιλάμε για αερομεταφορείς οι οποίοι είναι απολύτως υπεύθυνοι για τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν απέναντι στους επιβάτες. Και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση κάποιοι αερομεταφορείς να είναι υπεύθυνοι για αρνητικές καταστάσεις τις οποίες έχει βρεθεί ο ίδιος ο επιβάτης ή η αποσκευή του επιβάτη για το οποίο δεν έχει καμία σχέση όμως η επιχείρηση. και θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση ο αερομεταφορέας να ζητήσει αποζημίωση από κάποιον τρίτο. Σαν παράδειγμα, όταν ξεφορτώνει κανείς ε, τα πράγματά του με τις υπηρεσίες εδάφους και πάθουν κάποια ζημιά, ε, φταίνε οι υπηρεσίες εδάφους, αλλά ο επιβάτης δεν τον ενδιαφέρει, θέλει να αποζημιωθεί γρήγορα και η αποζημίωση θα πρέπει να δοθεί από την εταιρεία, την αεροπορική, γιατί αυτή είναι σε επαφή με τον πελάτη και η εταιρεία θα πρέπει να είναι πλέον σε θέση να ζητήσει την επιστροφή των δαπανών της αυτών από τις εταιρείε υπηρεσιών εδάφους που προκάλεσαν τη ζημία. Πέμπτον, σχετικά με το 1107 το 2006 κανονισμό. Νομίζω ότι σαν ρύθμιση δεν είναι κακή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί σωστά. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι με περιορισμένη κινητικότητα και οι ανάπηροι έχουν ε, προβλήματα και στα αεροδρόμια, στις μετακινήσεις τους στα αεροδρόμια. Είναι επίσης γνωστό ότι κάποιες επιχειρήσεις ζητούν επιπλέον χρήματα για το μέσο μετακίνησης ή για τον εξοπλισμό τον οποίο παρέχουν. Έχω συζητήσει το θέμα αυτό επανειλημμένα Έχω συζητήσει επίσης ε, και το θέμα των γονέων που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους μόνοι τους. Θα πρέπει οι μετακινήσεις των παιδιών να διευκρινιστούν καλύτερα και οι γονείς οι οποίοι ε, ταξιδεύουν με τα παιδιά τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Όπως είπα λοιπόν από πριν, συμφωνώ με κάποιες από τις προτάσεις του εισηγητή, αλλά έχω και ορισμένα προβλήματα. Στο άρθρο 6, οι επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση βέβαια να είναι ενήμερη σχετικά με τα δεδομένα PNR, τα οποία έχει στη διάθεσή του αερομεταφορέας. Αλλά ο εισηγητής πηγαίνει ακόμα παραπέρα και λέει ότι δεν θα πρέπει να αρνούμεθα στους επιβάτες την είσοδό του στο αεροσκάφος επί τη βάση των δεδομένων PNR εκτός και αν είναι ύποπτη τρομοκρατικών ενεργειών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ γιατί πολλές φορές ε, η τρίτη χώρα ερμηνεύει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με το PNR και ταυτόχρονα ο επιβάτης θα πρέπει να διορθώσει τα λάθη τα οποία έχουν γίνει κατά τη διάρκεια <clears throat> της κράτησης. Αν έχω γράψει λάθος το όνομά μου σαν παράδειγμα ή αν έχω βάλει λάθος ημερομηνία γέννησης, τότε το ειστήριό μου απλά δεν είναι έγκυρο. Το πρόβλημα είναι ότι αν εμείς δίνουμε 48 ώρες δυνατότητα να αποσυρθεί μια κράτηση, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί η τιμή της κράτησης του εισιτηρίου εξαρτάται από τη στιγμή της αγοράς. Υπάρχει όμως η δυνατότητα μέσα σε δύο ώρες να υπάρξει ανάκληση της κράτησης. Έχω επίσης αμφιβολίες για την ανάγκη να πετάει κανείς προς μία κατεύθυνση έτσι ώστε να μπορέσει να αγοράσει και το εισιτήριο της επιστροφής και έχω επίσης πρόβλημα και με το θέσφατο το οποίο ε, <clears throat> σημειώνει ο εισηγητής σχετικά με την αγορά εισιτηρίων προς, ε, τρίτους, προς τρίτα πρόσωπα. Μερικές φορές ε, μέσα στο χρόνο τα εισιτήρια, ας πούμε τώρα πριν τις γιορτές, είναι πιο ακριβά και κάποιοι κερδοσκόποι θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα εισιτήρια εκ των προτέρων για να μπορέσουν να τα ξαναπουλήσουν και να κερδίσουν χρήματα συμφωνώ ότι θα πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του επιβάτη με κάποια χρέωση βέβαια. Και ένα άλλο θέμα είναι το τι ε, στοιχεία PNR επηρεάζονται από τέτοιες αλλαγές. Τώρα, για τους επιβάτες που έχασαν τις ε, αποσκευές τους ή που καθυστερούν, δεν θα πρέπει να έχουν την ίδια αποζημίωση ε, για αυτούς οι οποίοι καθυστερούν ε, το ταξίδι τους. Εδώ έτσι και αλλιώ ανοίγει αν θέλετε χώρος για καταχρήσεις. Γιατί αν κάποιος για τη βαλίτσα του όταν τη χάσει θα μπορέσει να του πληρώσει το, η εταιρεία κάποιο φαγητό ή ε, μία νύχτα στο ξενοδοχείο, τότε θα αρχίσουν οι επιβάτες να χάνουν τις βαλίτσες τους για να τους πληρώνουν τζάμπα ξενοδοχείο. Λοιπόν, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος ε, των υπολείπων επιβατών και έτσι και αλλιώς θα καταθέσω αρκετές τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και εγώ νόμιζα ότι οι Ισπανοί ήταν αυτοί που μιλούσαν γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος. Ο Σάσολη για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τον εισηγητή, τον κύριο Τέιλορ, για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, διότι έχουμε τη δυνατότητα τους ε, επιβάτες στους επιβάτες να δώσουμε δυνατότητα να μάθουν τα δικαιώματά τους. Η έκθεση κατά την απόψή μου είναι ισόρροπη, είναι πολύ καλά δομημένη. Εγώ θα ήθελα απλά να εκφράσω κάποιες απόψεις δικές μου και να κάνω κάποιες ε, διευκρινήσεις, γιατί έχω καταθέσει και κάποιες ε, τροπολογίες. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος κύριος ε, Τέιλορ, ότι δηλαδή είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί αυτό το ποιε είναι οι έκτακτες, ειδικέ συνθήκες. Κάτι το οποίο είπε και ο εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Κοινωνικής Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους ε, επιβάτες ε, και ε, εφόσον λοιπόν τους βοηθήσουμε, αυτό θα συνδράμε, θα συμβάλλει στο να εξευρεθεί το συντομότερο δυνατόν μια λύση στη διάσταση των απόψεων. Έτσι λοιπόν ο επιβάτης θα μπορεί να αποζημιωθεί ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό είναι δικαίωμά του. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί λιγάκι και αυτό το θέμα το PNR, αυτός ο κατάλογος ε, με τα ονόματα των επιβατών. Ε, τι είδους στοιχεία καταχωρίζονται και τελικά πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί περιλαμβάνονται πάρα πολλά στοιχεία. Ο αριθμός της ψωτικής κάρτας, οι ε, διατροφικές προτιμήσεις, ε, τα θρησκευτικά πιστεύω. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς πρέπει να επιμείνουμε να καταχωρίζονται μόνο τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα στην αεροπορική εταιρεία για να κάνουν την κράταση, κράτηση για τον επιβάτη, ε, σεβόμενες όμως την ιδιωτική σφαίρα του επιβάτη. Ε, και πάλι λοιπόν σε σχέση με το PNR θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο κύριο Τέιλορ να διευκρινίσει λίγο το τελευταίο κομμάτι του 6 που λέει ότι δεν επιτρέπεται άρνηση επιβίβαση σε επιβάτη λόγω του PNR εκτός εάν υπάρχουν ειδικέ υποψίες περί τρομοκρατίας στην ε, περίπτωση αυτή, ε, αν κάποιος είναι ύποπτος για ε, τρομοκρατικές πράξεις, νομίζω ότι πλέον αυτό είναι θέμα αστυνομίας και δεν είναι θέμα αεροπορικής εταιρεία, γιατί αν το κάνει αυτό η αεροπορική εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Η ασφάλεια λοιπόν του επιβάτη θα πρέπει να διασφαλίζεται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, αυτό το οποίο μπορούν να προσφέρουν όμως οι αρμόδιες εταιρείε ή υπηρεσίε. Και κάτι άλλο. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφάνεια στι τιμέ. Γιατί πάρα πολύ συχνά, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά και εμεί οι βουλευτέ, πολύ συχνά λοιπόν βλέπουμε ότι η τιμή που διαφημίζεται ιδιαίτερα από τις low cost εταιρείες δεν έχει καμία σχέση με την τελική τιμή του εισιτηρίου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει λοιπόν να εγγυόμεθα ότι οι τιμές που αναφέρονται για το εισιτήριο να είναι δικαιολογημένες οι τιμές. Δεν είναι δυνατόν να αγοράζει κανείς online ένα εισιτήριο και κατόπιν να διαπιστώνει ότι οτιδήποτε προστίθεται, ε, οτιδήποτε προκύπτει προστίθεται στο εισιτήριο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι επίσης απαράδεκτο το κόστος ε, του εισιτηρίου να επιβαρύνεται και από ένα συντελεστή που να έχει σχέση με την οδηγία, ε, με το κανονισμό αυτό που συζητάμε. Πρέπει λοιπόν να μπορεί επίσης να αποζημιώνεται ο επιβάτης όταν υπάρχει καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης. Η εταιρεία είναι εκείνη που αποζημιώνει. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ε, διότι οι υπόλοιποι πληρώνουν αυτό που θα έπρεπε να λάβει ο επιβάτης ως αποζημίωση. Και κάτι άλλο, η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι καθοριστική σημασίας, κυρίως όταν μιλάμε για μικρά παιδιά για μωρά, αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή ένα παιδί που μπαίνει στο αεροπλάνο κάτω της ηλικίας ε, των δύο ετών ταξιδεύει στην αγκαλιά της μαμάς ή του μπαμπά. Και Εάν έχουμε όμως δύο παιδιά, το ένα παιδί το δίνουμε σε ένα τρίτο επιβάτη, άγνωστο. Λυπάμαι, αλλά αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Ε, και το μωρό έχει δικαίωμα να ταξιδεύει με ασφάλεια. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι σωστό στα αεροπλάνα μέσα να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ασφαλή θέση, κάθισμα σε επιβάτη, ακόμα και πολύ μικρό και σε μωρό. Να προσφέρουν καροτσάκια, όπως αυτά που βάζουν σε αυτοκίνητα. Να κάθονται εκεί τα μωρά. Ε, κατά τα άλλα, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Αντιμετωπίζουμε εδώ μια μεγάλη οικονομική κρίση. Πρέπει λοιπόν να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες ε, των οικογενειών. Ε, το να ε, προσφέρει κανείς το ίμιση του εισιτηρίου σε παιδιά μέχρι της ηλικία των 5 ετών, αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανάγκες των οικογενειών. Και μια τελευταία παρατήρηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι οι επιβάτες που έχουν χάσει τις αποσκευές τους ή φτάνουν καθυστερημένα οι ε, αποσκευές αυτές, οι επιβάτες αυτοί πρέπει να αποζημιώνονται ακριβώς όπως και εκείνοι οι άλλοι επιβάτες που υπέστησαν καθυστέρηση. Τώρα, αν η εταιρεία δεν ε, ε, αντιμετωπίζει σωστά και γρήγορα το θέμα των αποσκευών, αυτό είναι λάθος ε, και η εταιρεία ε, θα πρέπει λοιπόν να αποζημιώσει τον επιβάτη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, αρχίζω να χάνω την υπομονή μου ζητώντας σας να είσαστε στην ώρα σας. Γι' αυτό λοιπόν αυτή είναι η τελευταία μου έκκληση που κάνω. Η κυρία Γκρίσμπεργκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Πράγματι να σεβαστώ το χρόνο αλλά δεν ξέρω ποιο χρόνο. Δύο λεπτά, δέκα λεπτά, πέντε λεπτά, εφτά λεπτά. Πέντε, πέντε, πέντε. Α, ωραία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα πω σε πέντε λεπτά σύντομα. <clears throat> Να ευχαριστήσω λοιπόν εγώ τον Κιθ Taylor για τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, τις οποίες βρήκα πάρα πολύ χρήσιμες. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω και ό,τι δεν προλάβω να πω θα το διατυπώσω μέσα από τις τροπολογίες μου στο κείμενο του Τέιλορ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μας είπανε πολύ, όπως και η ΟΚΕ, οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ, είναι σαφής, έχει διευκρινιστεί από την ομολογία και εγγράφει ένα πλαίσιο ευθυνών σαφές θεωρητικά. Στην πραγματικότητα, η έκθεση αυτή έρχεται σε σωστό χρόνο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάπως καλύτερα και σε σχέση με τα δικαιώματα και σε σχέση με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών. Δεν θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο Keith Taylor για την ενημέρωση των επιβατών για τα δικαιώματα τους, γιατί διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ κατανοητά από όλου. Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι απαραίτητο να έχουν όλη την ίδια ενημέρωση μέσω ενός σαφούς συντόμου εγχειριδίου. Τώρα για τις τηλεφωνικές επαφές, ιδιαίτερα για τις low cost εταιρείε, όπου οι επιβάτες δεν έχουν καμία δυνατότητα επαφής, διότι δεν υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία για αυτούς όταν έχουν προβλήματα. Σχετικά με τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο είναι ένα σημαντικότατο δικαίωμα και γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί με σωστό τρόπο. Υπάρχει ένα μικρό στοιχείο το οποίο μου διαφεύγει και το οποίο ίσως οι μεν και οι δεν θα μπορέσουν να μου διευκρινίσουν. Ε, ναι μεν συμφωνώ με τον ε, μη μεταφερόμενο χαρακτήρα των εισιτηρίων, το ότι ο επιβάτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το αλέ για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την επιστροφή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ένας επιβάτης ο οποίος πήγε σε ένα μέρος με μια άλλη πτήση ή με ένα άλλο μέσο για διάφορους λόγους να μην μπορέσει να χρησιμοποιήσει το εισιτήριο της επιστροφής του. Αυτό ίσως είναι μια μικρή λεπτομέρεια αλλά έχει μεγάλη σημασία για τους επιβάτες και πρέπει να διευκρινιστεί. Σχετικά τώρα με την ισορρόπηση των διαφόρων συμφερόντων, προφανώς και εγώ θα ήθελα να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση απώλειας μιας αποσκευής και της πιθανής αποζημίωσης. <clears throat> Αυτό είναι κάτι που θίγει εκατομμύρια επιβατών στην Ευρώπη. Αν τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των αποσκευών φτάνει στο στόχο τους, ε, κάποια δεν φτάνουν ποτέ. Και εδώ δεν θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Κέιτ, Κίθ, γιατί προτείνει οι επιβάτες των οποίων έχουν καθυστερήσει οι αποσκευές να πάρουν σαν αποζημίωση ακριβώς την αποζημίωση που παίρνουν οι καθυστερημένοι επιβάτες. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία εδώ και σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες των αερομεταφορέων, ανάμεσα στην απώλεια μιας εποσκευής η οποία θα πρέπει να τύχει αποζημίωσης και στις δυσκολίες που οδηγούν στην καθυστέρηση ενός επιβάτη. Θα πρέπει να βρούμε, θα έλεγα, μια κάποια αναλογικότητα εδώ σε σχέση με την αποζημίωση. Τώρα, για τα PNR. Νομίζω ότι όπως είπε και ο ε, εισηγητής ότι θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα για λόγους ισορροπίας θα έλεγα να είμαστε ενήμεροι για τα PNR, τα προσωπικά που μας κρατούν οι αερομεταφορείς και οι επιβάτες δεν θα πρέπει να τους αρνούνται την είσοδο στο αεροσκάφος λόγω του φακέλου τους, εκτός αν η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές. Και θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές, οι αστυνομικές αρχές, οι αρχές ασφαλείας να διαχειρίζονται πιθανώς την απόρριψη ενός επιβάτη ή να ζητούν από τον επιβάτη αυτό να φύγει από το αεροπλάνο την τελευταία στιγμή. Κάτι τέτοιο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουν οι αστυνομικές αρχές, οι αρχές ασφαλείας και ουχή αερομεταφορής. Και τέλος κλείνω για το 11.07 του 06 για τα PNR πάλι. Νομίζω για όλους τους Ευρωπαίους είναι απαράδεκτο τα πρόσωπα αυτά να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους επιβάτες η άρνηση ε, να μπει ε, ένας ε, επιβάτης με περιορισμένες δυνατότητες κίνησης στο αεροσκάφος είναι από μια άλλη εποχή, είναι κάτι το πάρα πολύ ξεπερασμένο. Κάποιες εταιρείες πράγματι ασκούν διακρίσεις αρνούμενοι τους αναστούς αναπήρους την είσοδο στο αεροπλάνο για λόγους υποτίθεται ασφαλείας. Οι low cost το κάνουν αυτό που θέλουν να μειώσουν το κόστος εκμετάλλευσης και δυστυχώς ασκούν διακρίσεις. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει η βοήθεια που θα δίδεται στα πρόσωπα αυτά να είναι σαφής και ξεκάθαρη τη στιγμή που κρατούν το εισιτήριό τους. Το ίδιο και για τις βαλίτσες τους. Τώρα, για τις βαλίτσες ακριβώς αυτών των ανθρώπων περιορισμένης κινητικότητας, Ξέρω ότι μιλάω γρήγορα, αλλά κάθε ζημία η οποία προκαλείται σε ένα μέσο κίνησης θα πρέπει να αποζημιώνεται πλήρως, διότι δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς τη χρησιμότητα αυτών των μέσων μετακίνησης με τις βαλίτσες, γιατί τα μηχανήματα και οι εξοπλισμοί μετακίνησης είναι απόλυτα απαραίτητοι για την κίνησή τους. Ευχαριστώ, κυρία Γκρισμπέκ. Αυτό το παράδειγμα ήταν τρομερό. Όλοι καταλάβαμε τι μπορεί κανείς να πει σε πέντε λεπτά. Τα πάντα δηλαδή. Η κυρία Φώστερ. Εδώ νομίζω ότι θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι, Τζάκι. Okay, um, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε κάποια σημεία. Γιατί ο λόγος που πιστεύω ότι ξανακοιτάμε τους κανονισμούς αυτούς συχνά έχει να κάνει με την κατάσταση που είχαμε με το ηφαίστειο της Ισλανδίας πέρυσι και τις ε, δικαστικές αποφάσεις στη συνέχεια. Οπότε για μένα από εκεί απορρέει η ανάγκη για αλλαγέ. Γι' αυτό λέει η Επιτροπή ότι πρέπει να τους κοιτάξουμε αυτούς τους κανονισμούς. Πολλά πράγματα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στους αρχικούς κανονισμούς. Εδώ στην Επιτροπή μας, ε, Πρόεδρε, ε, φροντίσαμε για αυτούς και πολλά από αυτά ισχύουν ακόμα. Νομίζω ότι οι αρχικοί κανονισμοί ήταν πάρα πολύ καλοί. Εννοείται, τόσο περνά ο καιρός, πρέπει κανείς να βλέπει πώς μπορεί να διευκρινίσει ακόμα περισσότερο κάποια στοιχεία τους. Έχουμε μια ανησυχία, όπως είπε και ο συγητής, η συνεδριάσαμε και είπε ότι έλαβε υπόψη του αυτά που είπαμε εμείς. Όμως, το κείμενο που είχε πριν από εκείνη τη συνάντηση και το κείμενο ε, στο οποίο κατέληξε μετά τη συνάντηση είναι ίδια όλος περιόργος. Οπότε δεν καταλαβαίνω ότι μια μισή ώρα που συνεδριάσαμε τι έλαβε υπόψη του. Τίποτα από ό,τι φαίνεται, αλλά έτσι κι είναι δικό του θέμα, εκείνος θα αποφασίσει. Δύο πράγματα. Ποιες είναι οι έκτακτες περιστάσεις. Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Άλλο είναι ε, ανωτέρα βία και άλλο είναι οι έκτακτες περιστάσεις. Οι έκτακτες ε, περιστάσεις και η ανωτέρα βία είναι κάτι το οποίο νομικά διευκρινίζεται. Αλλά αν αρχίσεις να κάνεις έναν κατάλογο, από πού ξεκινάς και πού σταματάς. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο το, στο 295, έτσι κι αλλιώς έχει να κάνει με τη σύμβαση του Μόντρελ, έτσι, είναι καλά γραμμένο. Ίσως να έχει αλλάξει λίγο, αλλά γενικά και το 14 και το 15 το αρχικό κειμένου είναι καλά. Στη συνέχεια τώρα, άμα πάμε πιο πέρα, το 6 και το 7 για τα PNR. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάζει άλλος κανονισμός. Δεν πρέπει εδώ να μπούμε στο PNR. Δεν βλέπω ότι θα μπορούσε κανείς να πει εδώ. Επίσης για το θέμα της πτώχευσης. Θυμόσαστε τι συζήτηση είχαμε στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και εδώ ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς θα χειριστούν το θέμα με διάφορες εταιρείες στην περίπτωση που έχουμε τέτοιες περιστάσεις. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας το διευκρινίσει. για το θέμα των εισιτηρίων. Όπως και ο συνάδελφος Κρίσμπερκ, έτσι και εγώ πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο σας λένε ότι ε, τα, τα εισιτήριά σας ε, ακυρώνονται αν δεν εμφανιστείτε, είναι γιατί αλλιώς θα τους μείνει καινή θέση. Είναι δηλαδή εμπορικές πρακτικές Αλλιώς μπορούμε να αγοράσουμε one-way εισιτήριο. Είναι εμπορικέ οι αποφάσει αυτέ. Τώρα για την ε, αλλαγή του ονόματο, πώ δηλαδή μεταφέρεται το εισιτήριο από τον ένα στον άλλον, τον έφερα και κάποιοι. Ε, κοιτάξτε. Μα έτσι μεταφτάνουμε στο PNR. Ο η συγητής μιλάει για τις αποζημιώσεις. Μα ήταν πάρα πολύ δύσκολο έτσι καλλιώς να φτάσουμε στις αποζημιώσεις που φτάσαμε. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε. Είναι αδύνατο, ήταν εφιάλτης να καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε. Πού να ξανανοίξει το θέμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξανανοίξει το θέμα αυτό. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τα αφήσουμε. Έπειτα, το θέμα της ε, βοήθειας. Ε, Κάποιος είχε πάει στα Βαρμπέντο σε ένα ξενοδοχείο και μετά από εκεί ε, ήθελε να κάνει μια προσφυγή. Πρέπει να προσέξουμε πολύ τελικά τι θέλει να κάνει κανείς. Αργότερα θα σας πω και το όνομα, αν με κοιτάτε έτσι. Θα σας πω ποιος ήταν. Η αλλαγή του ονόματος. Ναι, μπορεί κάποιος να κάνει ένα λάθος, αλλά 48 ώρες δεν νομίζω, γιατί όντως οι τιμές αλλάζουν. Πάλι είναι εμπορικό το θέμα εδώ και για τις αποσκευές πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τη σύμβαση του Μόντρεαλ. Τα επίπεδα αποζημίωση δηλαδή αναφέρονται εκεί ποια είναι η αποζημίωση για απώλεια αποσκευής. Αν κάποιοι αερομεταφορείς ε, δίνουν περισσότερα, βασικά εμένα μια φορά μου καταστρέψανε τη βαλίτσα και μου δώσανε μια καινούρια για τα PRM, που είναι τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Μιλήσαμε γι' αυτό και στην συνάντηση που είχαμε. Η πρόσβαση τους είναι φυσικά δωρεάν, υπάρχει οξυγόνο, υπάρχουν όλα, αλλά αν κάποιος Ορισμένοι χρειάζονται 24 ώρες οξυγόνο και έχουν δικέ τους συσκευές. Το θέμα είναι οι δικές τους συσκευές ότι πρέπει να προσαρμόζονται στις ασφαλείς προδιαγραφές. Αυτό όντως πρέπει να συζητηθεί. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, γιατί όλα εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο επιβάτης που έχει ανάγκη από τον εξοπλισμό αυτό υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε έναν επιβάτη που μπορεί να περπατήσει και σε έναν που δεν μπορεί να περπατήσει. Αν πρέπει να φέρει και την ε, ε αναπηρική του πολυθρόνα είναι αλλιώ από ότι αν δεν τη χρειάζεται. Για τα παιδιά τώρα που λέγατε για τα μωρά, είναι κάτι διαφορετικό από τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα υπάρχουν κανόνες νομικά. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα μωρά, απλώς προσοχή πώς αντιμετωπίζετε την κάθε περίπτωση και τι γλώσσα χρησιμοποιείτε για κάθε περίπτωση. Εδώ πέρα μιλάμε για διεθνείς μεταφορές, έτσι, τις αεροπορικές. Τέλος, πολλά από αυτά που λέει ο συγητής ε, δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Ένα-δυο πραγματάκια, ναι, με βρίσκουν σύμφωνοι. Η ατζέντα του συγητή δεν με βρίσκει σύμφωνη δεν έχει τίποτα να κάνει αυτά που προτείνει δηλαδή ο συγητής, με το λόγο για τον οποίο θελήσαμε να ξανακοιτάξουμε τους κανονισμούς αυτούς. Γι' αυτό και θα υποβάλω διάφορες τροπολογίες και τα μέλη της Επιτροπής αυτής Εντάξει, είναι εύκολο να τα θέλουμε όλα ωραία και καλά, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να διευκρινίζουμε ε, τα πράγματα τα οποία χρειάζονται πραγματικά αλλαγές. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Μάικλ, ε, θα έρθουμε και σε σένα εντό λίγου. Νομίζω ότι είσαι επόμενο. Ο κύριο Κόπ. για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον κύριο Τέλερ για το σχέδιο της έκθεσης. Έχω τρεις ε, παρατηρήσεις. Πρόκειται για ένα γενικότερο πρόβλημα της εποχής μας. Είναι αληθές και σωστό ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά κάπου αναφέρεται ότι υπάρχουν και υποχρώσεις. Όποιος ταξιδεύει με το αεροσκάφος ε, πρέπει και ο ίδιος να συμβάλλει έτσι ώστε το ταξίδι να είναι ασφαλές. Και κάπου πρέπει να εμφανίζεται αυτό. Δεύτερον, ο κανονισμός για τα δικαιώματα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό. Εμένα με ενδιαφέρει ε, τελικά ποιος φταίει. Γιατί και οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και τα αεροδρόμια έχουν ε, και οι δύο συμβάλλει στο να μην εφαρμόζει αυτό που εγκρίναμε πριν από πέντε χρόνια. Και ένα τρίτο σημείο. Έχω δει μου, μόνος μου ότι οι άνθρωποι ε, με πρόσθετα μέλη από μέταλλο υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Ε, ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, ένα πρότυπο, έτσι ώστε να υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση. Ίσως ε, κύριε Τέιλορ μπορούμε λιγάκι να καλέσουμε την Κομισιόν να ε, διεκδικήσει, να θελήσει να εισάγει ένα κοινό διαβατήριο πρόσθετων μελών. Ε, καταρχήν λοιπόν ε, τα δικαιώματα των επιβατών δεν υπάρχουν για να εφαρμόζονται συχνά και για να ε, εκτιναχθούν οι τιμές γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αλλά εμείς επιθυμούμε τα δικαιώματα των επιβατών να μην τίθενται συχνά επιτάπητος, ε, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι αεροπορικές εταιρείε να μην μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Και τι συμβαίνει συχνά, ακούμε ένα αεροσκάφος ε, να έχει καθυστέρηση γιατί υποτίθεται ότι έφτασε αργά στο αεροδρόμιο. Γιατί είναι ε, τόσο τσιμα-τσιμα όλα αυτά τα ωράρια. Και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ε, κατ' ουσίαν κόλαφος για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είπαμε ε, να υπάρχει αποδεικτή καθυστέρηση μέχρι και πέντε ώρες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε απαράδεικτο μετά από τρεις ώρες το πολύ πολύ. Εμείς ε, λοιπόν στις αεροπορικές μεταφορές ε, δεν χειριζόμαστε τα πράγματα σωστά και λέμε και ζητάμε μια ανεξάρτητη υπηρεσία διαιτησίας. Πέταγα από τη Σόφια στη Βιέννη έξι ώρες ε, καθυστέρηση γιατί ποτέ χιόνισε στη Βιέννη λες και δεν είχε ξαναχιονίσει. κάποια στιγμή έκλεισε το αεροδρόμιο. Εγώ όμως είχα πέντε ώρες καθυστέρηση και η αεροπορική εταιρεία μου είπε θα σας δώσω 25 ευρώ. Μα αυτό ήταν γελίο. Έφτασα στη Βιέννη στι 2 η ώρα το βράδυ και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει λοιπόν ανεξάρτητη αρχή διαστησία και επειδή δεν υπάρχει αυτή και δεν αντιδρούν και ευρωπαϊκέ εταιρείε, μπορεί κανεί να απευθυνθεί ε, σε έναν ιδιώτη δικηγόρο. Αν κερδίσει τη δίκη θα πάρει το 20% ε, αλλά κανονικά θα έπρεπε να έχουμε μία ανεξάρτητη ε, αρχή διαιτησίας. Και τώρα έχω αυτή τη ε, διαμάχη με την Air Berlin, οι οποίοι όμως ε, δεν ε, λένε τίποτα, περιμένουν μέχρι να φτάσουν τα πράγματα στο απροχώρητο και μετά καταλήγουν σε κάποια συμφωνία με το δικηγόρο. Αυτό όμως δεν γίνεται όλη αυτή η καθυστέρηση. Ζούμε σε κράτος δικαίου και δεν είναι δυνατόν να πρέπει εγώ να γράψω τρεις-τέσσερις φορές για να δικαιωθώ. Στις συνδρομικές μεταφορές φορές ε, υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή ε, διαιτησίας, ξέρουν πότε ε, μπορώ να δικαιωθώ και πότε όχι. Όμως στις αεροπορικές μεταφορές στο 99% των περιπτώσεων πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος επιβάτης και γι' αυτό πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Μετά, όταν γίνονται διορθώσεις λόγω λάθους, γράψαμε, ας πούμε έγραψα λάθος το όνομά μου ή ε, την ημερομηνία γέννησής μου και το άλλαξα μετά από δύο ώρες ε, και μου λέτε να πληρώσω, μα δεν είναι δυνατόν αυτό. Και όσον αφορά το αλέ ρετούρ, βεβαίως ε, και το ρετούρ θα μπορούσε να απαγορευτεί. Όμως, αν έχουμε χρησιμοποιήσει το αλέ, μπορούμε να ξεχάσουμε το ρετούρ, γιατί έτσι το έχουμε βγάλει μόνο και μόνο για να πέσει η τιμή. Αν όμως ε, δεν πάω στο ρετούρ, πάλι είναι ελεύθερη θέση. Πού είναι η διαφορά. Όλα αυτά είναι εις βάρος των επιβατών. Ο ανώτατος άρχον είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Και δεν μπορούμε να έχουμε πάλι μια απόφαση που θα λέει ότι πρόκειται για αθέμητον ανταγωνισμό. Εμείς ε, χρειαζόμαστε δίκαιους ε, κανόνες για όλους. Είτε όλοι με αποζημίωση μετά από μία ώρα ή κανένας. Αυτό δεν είναι επικουρικότητα, είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Κατόπιν τούτου είτε ευρωπαϊκός κανονισμός για όλους ή για κανένα. Είναι λοιπόν σωστό να αναθεωρηθεί το θέμα, αλλά εξακολουθούμε να απέχουμε πόρο από όλα αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ο κύριος Higgins, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Θα δω τι μπορώ να πω σε πέντε λεπτά. Υπάρχουν, θα έλεγα, σημεία της έκθεσης που είναι καλά, αλλά ίσως υπερβάλλει λίγο η συγητής σε σχέση με την ισορροπία των συμφερόντων του ε, καταναλωτή, επιβάτη και της εταιρείας. Συμφωνώ με τη Φώστερ ότι έχουμε καταλήξει σε μια ισορροπημένη σχέση σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και έχουμε ξεφύγει από τα απαράδεκτα φαινόμενα που ζούσαμε στο παρελθόν. Η 8, παράγραφος 8, θετική, καλύτερη ενημέρωση. Ε, παράγραφος 5, είναι ζωτικό να υπάρχει περισσότερο προσωπικό όταν αναβάλλεται ή καταργείται μία πτήση που αφήνουν τους επιβάτες μόνους. Ξέρετε τι γίνεται με εταιρείε όπως η Ryanair σχετικά με την πιθανή επιβάρυνση την οποία πληρώνει, καλείται να πληρώσει ο επιβάτης, έχουν εφεύρει όλων των ειδών της επιβαρύστης προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι σαφές επίσης ότι οι 48 ώρες για τη διόρθωση ενός λάθους είναι κάτι το πάρα πολύ υπερβολικό. Πρέπει μέσα σε δύο ώρες να υπάρξει η, η διόρθωση. Συγγνώμη. Τώρα για την παράγραφο 18, για την αποζημίωση για τις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να αποζημιώνουμε για τις καθυστερημένες αποσκευές με τον ίδιο τρόπο που αποζημιώνουμε για τους καθυστερημένους επιβάτες. Επίσης οι επιβάτες όταν θέλουν να κάνουν μια διαδικασία επαφής ή να ζητήσουν μια αποζημίωση μπορούν να το κάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το 22 είναι προβληματικό, δεν είναι ρεαλιστικό, πρέπει να αποσύρει την πρόταση αυτή ο εισηγητής. Και η 30 είναι καλή πρόταση, ιδιαίτερα για τους επιβάτες περιορισμένης κινητικότητας. Κάτι το οποίο θέλω επίσης να υπογραμμίσω είναι ότι τα ίδια δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές μεταφορών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το επιβάλλουμε ε, στις λεωφοριακές γραμμές. Άλλο τα αεροπλάνα, άλλο τα λεωφορεία. Ευχαριστώ κύριε Χίγγινς και εγώ θα ήθελα λίγα λεπτά και ε, κυρία Γκρίσμπεκ θα με ελέγξει αν ξεπεράσω το πεντάλεπτο. Πρώτον, θεωρώ ότι θα πρέπει να εγγράψουμε στην ομοθεσία κάποιες νέες ρυθμίσεις. Τα μέσα ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας θα γράψουν αυτά που λέω. Κάθε εταιρεία που λέει ότι θα πρέπει για λειτουργικούς λόγους να ανακοινώνει καθυστέρηση θα πρέπει ε, να ε, ε, τους επιβάλλουν ένα πρόστιμο το οποίο μπορεί να φτάνει εκατομμύρια κάθε φορά που χρησιμοποιούν αυτή την απαράδεκτη εξήγηση. Ε, καθυστέρηση λόγω λειτουργικών εν πάση περιπτώσει αιτιών. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, θα πρέπει να ζητήσουμε από τις εταιρείες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτήν τη σαχλαμάρα όταν έχουν καθυστερήσεις θα πρέπει να δούμε τον κανονισμό αυτό με διαφορετικό τρόπο. Κάποια στοιχεία του κανονισμού είναι καλά, κάποια άλλα στοιχεία δουλεύουν ακόμα και τώρα σχετικά καλά. Από την άλλη όμως υπάρχουν σημεία του κανονισμού ενισχύ που δεν είναι πλέον λειτουργικά. Και όπως είπε και ο κύριος Χίγκινς, αναφέρθηκε σε μια εταιρεία της χώρας του, υπάρχουν εταιρείε που κάνουν ό,τι μπορούν να φορτώνουν τους επιβάτες μέσω της παραβίασης αυτού του κανονισμού. Και το κάνουν αυτό γιατί οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε καμία περίπτωση δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ έχω έναν εκλογέα ο οποίος ε, έχει καταθέσει μία μήνυση εναντίον της KLM. Ονοματίζω την εταιρεία. Χρησιμοποίησε και την ε, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας στη Μεγάλη Βρετανία και δεν βρήκε το δίκιο του ε, δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα. Η ΚΕΛΕΜ δεν απάντησε στον ε, εκλογέα μου, αλλά η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας μου είπε σκοτιστήκαμε, δεν είναι δική μας δουλειά. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να δούμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ομπουτσμαν για τις αερομεταφορές, κάποιον ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει, να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Ε, τώρα αυτές τις ε, περιφερειακές επιβαρύνσεις υπάρχουν κάποιες εταιρείες, στρέφομαι στον κύριο Higgins, που τους ε, ζητούν χρήματα από τους επιβάτες για να καταθέσουν την αίτηση αποζημίωσης. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι γίνεται σχετικά με το δικαίωμα της επιστροφής. Τι γίνεται με το φόρο τον οποίο πληρώνουν οι ε, επιβάτες ε, όταν δεν μπορούν να πετάξουν επειδή είναι άρρωστοι κτλ. Και όταν προσπαθούν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους συστηματικά το κόστος ε, το οποίο ε, ε, κοστίζει ακριβώς η προσπάθεια που κάνουν για να πάρουν τα λεφτά πίσω, η διαδικασία έχει τέτοιο κόστος το οποίο είναι συστηματικά μεγαλύτερο από το κόστος του εισιτηρίου. Λοιπόν, ενώ θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να επιστρέφονται, Σορεύονται λοιπόν χρήματα, κερδίζουν χρήματα απαράδεκτα. Λοιπόν, η κυρία Φώστερ έχει δίκιο βέβαια ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια της ισχύουσας νομοθεσίας που είναι καλά. Οπότε ας τα κρατήσουμε αυτά και ας προσπαθήσουμε να τα διατηρήσουμε. Υπάρχει θέμα και με τη χρονική προθεσμία. Σαν παράδειγμα όταν έχουμε ας πούμε την ηφαιστειακή τέφρα. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα στις αερομεταφορές από ό,τι κάνουμε στις μεταφορές και στις μεταφορές με Λοιπόν, α στείλουμε το μήνυμα στις αεροπορικέ επιχειρήσεις να πάψουν να μαζαλίζουν με την καθυστέρηση για λειτουργικούς λόγους, γιατί αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κυρία Γκρίσμπερ, τα κατάφερα. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση και τιμή για μας που μπορέσαμε να σας ε, ακούσουμε. Εξάλλου και το δικαστήριο σας άκουσε και στην υπόθεση 1 αποφάσισε ότι οι τεχνικές ε, προϋποθέσεις δεν είναι έκτακτες περιστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν χαίρεται για την πρωτοβουλία και για την έκθεση του κυρίου Τέιλορ και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πολύ για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε μαζί του. Η έκθεσή του είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Οι ενέργειες μεταφορές είναι το πρώτο είδος μεταφορών που προστατεύει τους επιβάτες. Έχουν επιτευχθεί πολλά, ε, νομοθεσία έχει υιοθετηθεί έκτοτε και οι άλλες μορφές μεταφορών. Θέλω πάντως να σας πω ότι μαζί σας υιοθετήσαμε ε, δικαιώματα επιβατών και για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τις ενέργειες και τις οδικές. Χαιρόμαστε πολύ λοιπόν για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα, μια που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκρινε ανακοίνωση για τα δικαιώματα των επιβατών για όλες τις μορφές μεταφορών. Και εκεί αναφέρει ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία, ε, από τα οποία χαίρει ο επιβάτης κατά την μεταφορά του. Συγχρόνως, Προ ενημέρωσή σα, πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού 261 για τους επιβάτες ενεργείων μεταφορών και θα κάνουμε και έκθεση επιπτώσεων όσον αφορά την αναθεώρηση αυτή του κανονισμού. Χαίρομαι από την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε για να ε, και υποφελούμε από αυτήν για να ζητήσω από όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην ανοιχτή αυτή διαβούλευση που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση που υπάρξουν τα κυρώσεις είτε καθυστερήσεις, είτε προβλήματα με τις αποσκευές τους κλπ. κλπ. Τι μέτρα δηλαδή θα έπρεπε να υιοθετηθούν για να βελτιωθεί η βοήθεια προς τον επιβάτη. Μετά την διαβούλευση θα ακολουθήσει η αναθεώρηση βάσει του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο του 2012. Συνεπώς κύριε Τέιλορ, κύριε Σίμψον και οι υπόλοιποι αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η έκθεσή σας και η έκθεση της ΟΚΕ φτάνουν την κατάλληλη στιγμή και αποτελούν μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην αυτή νομοθεσία. Επιτρέψτε μου βέβαια συγχρόνως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το σχέδιο έκθεση. Συμφωνούμε με τον καταναλωτή, με τον εισηγητή συγγνώμη, για το ότι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν όταν δεν υπάρχει συνοχή, όταν δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή στα κράτη-μέλη, όταν δεν υπάρχει σωστή νομική ερμηνεία και ίδια παντού ή το πρόβλημα της ε, αποζημίωσης. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει με την εκστρατεία ενημέρωσης και η κυρία Κούνεβα χτες άρχισε και πάλι τις επισκέψεις της ξεκινώντας από την Βαρσοβία υπέρ αυτής της εκστρατείας πληροφόρησης. Ξέρετε ότι έχουμε διάφορα πόστερ τα οποία κυκλοφορούν στα αεροδρόμια τα ευρωπαϊκά με το σκοπό αυτό. Αλλά και άλλες προτάσεις θα τις ακολουθήσουμε και στη συνέχεια με την ε, ε, αξιολόγηση επιπτώσεων θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση του επιβάτη, την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων του και τον ε, χειρισμό των ε, διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται. Για το θέμα της ε, πτώχευσης έχει ολοκληρωθεί μελέτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει τώρα τις αντιδράσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Είμαστε έτοιμοι πάντως να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μαζί σας για αυτό το θέμα. Τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με τη διαφάνεια των τιμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει έναν έλεγχο του, των ρυθμίσεων 2000, ε, το 2008 για να δούμε τι ισχύει στην αγορά και εφόσον δούμε ότι κάποια πράγματα είναι ξεπερασμένα θα τα διορθώσουμε. Πριν ολοκληρώσω όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι δουλεύουμε και πάνω σε ένα άλλο κείμενο για την ε, βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού 1107 για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή τα άτομα με αναπηρία. Είναι κάτι που θα υιοθετηθεί την άνοιξη του 2008 από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να είμαστε καλυμμένοι κατά την διάρκεια των παρολυμπιακών ε, αγώνων στο Λονδίνο και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα να μπορέσουν να αποφεληθούν. Κύριε Τέιλορ, αγαπητοί φίλοι της Επιτροπής Μεταφορών, εκ μέρους του επικεφαλής της ε, ε, μονάδας μας και εκ μέρους μου της Ιδίας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε μαζί σας. Θα αλλάξει το προσωπικό μας του χρόνου, ίσως θα τα διαβάσετε σε ένα press release. Όλοι πιστεύω τώρα στις διακοπές που έχουμε όλο και περισσότερες μετακινήσεις, ταξιδεύουμε πολύ, θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε εν ασφάλεια και θα επιστρέψουμε ωραία και καλά όλοι στις χώρες μας. Κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ. Κύριος Τέιλορ. Κύριος Τέιλορ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Δεν είναι υποχρεωτικό, άμα δεν θέλετε δεν πειράζει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους. Και περιμένω και τις τροπολογίες τις οποίες θα καταθέσετε. Κάτι μου λέει ότι θα καταθέσετε πολλές, αλλά εμπάσπερτο σοβαρά τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς να αποκλείουμε τίποτα θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τη βέλτιστη δυνατή λύση για τους επιβάτες και τα δικαιώματά τους. Αυτός είναι ο τίτλος. Δικαιώματα των επιβατών. Θα πρέπει λοιπόν εμείς τις υπηρεσίες που μπορούμε να διασφαλίσουμε από πλευρά των αερομεταφορέων να τις διασφαλίσουμε. Δεν είναι τόσο περίπλοκο. Περιμένω να εξετάσω όλες τις τροπολογίες σας και να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστώ κύριε Μπατάλια. Θέλετε να, προσθέσετε, να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχόμαι την ευκαιρία που μου δίνετε να σας εκθέσω κάποια θα έλεγα στοιχεία τα οποία μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι σημαντικά. Υπάρχουν θέματα τα οποία ίσως και δεν ακούστηκαν προηγουμένως, διαφάνεια σαν παράδειγμα, δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα στις διαφορετικές προσφορές, δυνατότητα για τον επιβάτη να επιλέξει. Αυτό δείχνουν ε, τα παράπονα των επιβατών, η έλλειψη επιλογής είναι ένα θέμα και πιστεύουμε ότι σε περιπτώσεις πτώχευσης ενός αερομεταφορέα εκεί αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη, καλύτερη διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω όλους, προθεσμία είναι η 12 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στη δεύτερη Ολομέλεια του μηνός Μαρτίου. Λοιπόν, 12 Ιανουαρίου προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Κλείνουμε την σημερινή και θα περάσουμε συνάντηση και περνάμε στους συντονιστές. Ευχαριστώ.